Καλησπέρα σε όλους. Ξεκινάμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Με το πρώτο σημείο στη μερίσια διάταξη, έχουμε στη μερήσια διάταξη τρία πιο σημαντικά σημεία, τις αναφορές για τα περιβαλλοντικά προβλήματα στην Ιταλία, κυρίως για την Καμπανία και το Φριούλι, ε, προβλήματα περιβαλλοντικά στην Ισπανία για ε, τους καπνούς και τις ε, εκπομπές στην Πολωνία. Στην Ισπανία είναι στην Γαλλικία. Η συζήτηση για την έκθεση πέτει για την, ε, το 2012 και η γνωμοδότηση του κύριου Τσίτσαστερ για τον εντοπισμό μιας θέσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν δύο αλλαγές στη μερίσια διάταξη που μοιράστηκαν στους συναδέλφους και αφορούν την έκθεση για τη Γαλλικία, για την αποστολή στη Ματρίτη δεν έχει ολοκληρωθεί διαπραγμάτευση για την έγκριση για αυτά τα δύο θέματα. Θα γίνει μια επιπλέον συζήτηση και η έγκριση θα λάβει χώρα στην επόμενη συνεδρία της Επιτροπής μας. Στις 5.30 θα σταματήσουμε τις εργασίες της Επιτροπής για να συνεδριάσουν συντονιστές. Επίσης υπάρχει και η έκθεση του, του κ. Σαλαβράκου για την, τον Ευρωπαίο Διαμεσολαβητή. Αν δεν υπάρχουν σχόλια, μπορείτε να υιοθετήσετε την τροποποιημένη πρόταση για την ημερήσια διάταξη. Επίσης, και σε αυτή την συνεδρίαση έχουμε μοιράσει στο παράτημα Β όλα τα θέματα που έχουν φτάσει στην Επιτροπή μας, τα οποία θεωρούνται μη σύμμορφα με τον καονισμό και επομένως δεν θεωρούνται παραδεκτά ε, δεν θεωρούνται παραδεκτέ αναφορέ. Τον κατάλογο αυτό όμω σα τον έχουμε μοιράσει και όπω συμφωνήσαμε με του συντονιστέ. εάν δεν υπάρχει αντίρρηση θεωρούμε ότι εγκρίνουμε την πρόταση όπω διατυπώθηκε. Με τον κατάλογο που έχει προσαρτηθεί και έχει μοιραστεί. Δεν υπάρχουν άλλε ανακοινώσει. Δεν βλέπω συναδέλφους που θέλουν την, το λόγο. Επομένως μπορούμε να περάσουμε στο πρώτο σημείο της ημερήσια διάταξης. Η έκθεση και η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για την διερευνητική επίσκεψη στην Πολωνία. Ο κύριος Μποστινάρου που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας θα πάρει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Επι... Ομολογώ ότι αυτή η διερευνητική τελευταία επίσκεψη που είχα την τιμή να οδηγήσω ήταν ίσως η πιο επιτυχής. Να σας πω γιατί. Καταρχήν οργανώθηκε με τρόπο εξαιρετικό και με αυτή την ευκαιρία εκφράζω την ευγνωμοσύνη και τις ευχαριστίες μας ε, προς τη Γραμματεία για το έργο της, εξαιρετικά οργανωμένο με εξαιρετική συνεργασία με το Γραφείο στο Βρότσλαφ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξαιρετικά χρονοδιαγράμματα για συναντήσεις με αναφέροντες και αρχές, Πολύ καλός χρόνος για να δούμε τους διάφορους συνομιλητές επιτόπου. Δεν υπήρξε ούτε ένα σημείο με ερωτηματικά για την οργάνωση. Δεν συμβαίνει συχνά να εκφράζουμε τέτοια ευγνωμοσύνη προς τη γραμματεία. Επιβάλλεται όμως και επιβάλλεται να εκφράσουμε τη βαθιά μας εκτίμηση για το έργο των David και Georgiana. Δεύτερον, υπήρξε εξαιρετική συνεργασία μεταξύ των Ευρωβουλευτών. Και αυτό δεν είναι σύνηθες. Είχα όμως την τιμή να συνεργαστώ με τον Κις Τέιλορ, από τον διακεκριμένο πράσινο συνάδελφο, και η ίδια ατμόσφαιρα και με τον ίδιο τρόπο όταν συνεργαστήκαμε με την κυρία Λίδια Ντεμπεργκ και τον κύριο Τσαρνέσκι, τον κύριο, τους, δύο, ε, τους δύο βουλευτές από τους Σοσιαλιστές Δημοκράτες και από το ECR αντίστοιχα. Η πρώτη εντύπωση ήταν ότι είχαμε αρκετό χρόνο για να ακούσουμε όλους τους αναφέροντες. Δεν υπήρξε ούτε ένας αναφέρον οργανωμένος ή μεμονωμένο πρόσωπο, ο οποίος δεν είχε το χρόνο να μιλήσει. Όλοι συζήτησαν μαζί μας, παρουσίασαν τα επιχειρήματά τους και εις επίμετρον είχαμε την τύχη να συναντήσουμε μια εξαιρετική οργάνωση από την πλευρά των αναφερόντων στην Λέντνιτσα οι οποίοι παρουσίασαν με powerpoints τα επιχειρήματά τους με τρόπο υποδειγματικό. Ήταν εντυπωσιακά καλή η παρουσίαση από άποψη τεχνική, από άποψη συνοχής, συνεκτικότητας, αλλά και από άποψη οργανωτική. Ήταν εξαιρετικά οργανωμένη και αυτό είναι ένα δείγμα οριμότητας και καλής οργάνωσης της κοινωνίας των πολιτών μέσα σε ένα κράτος μέλος. Επίσης σημαντικό ήταν ότι είχαμε αρκετό χρόνο για να ταξιδέψουμε και να δούμε χώρους που είχαν σημασία για τη δουλειά που πήγαμε να κάνουμε στην Πολωνία. Γιατί καμιά φορά μέσα από τα γυάλινα και αλουμινένια γραφεία μας βλέπουμε άλλη πραγματικότητα ε, από εκείνη που επικρατεί επί τόπου. Πάλι, να το ξαναπώ, ήταν εξαιρετική οργάνωση γιατί είδαμε τόπους, χώρους, προβλήματα και αποκομίσαμε ε, μια πρώτη ιδέα. Τέλος, όλα αυτά τα στοιχεία που ήθελα να σας παρουσιάσω ε, είναι ενσωματωμένα και ε, πραγματικά όλο τον υπερθετικό βαθμό χρησιμοποιώ αλλά είναι αλήθεια. Πρόκειται για εξαιρετικό σχέδιο έκθεσης της Τζορτζιάννα και νομίζω ότι με τη συμβολή των συμμετεχόντων, των ε, τακτικών μελών αλλά και άλλων θα έχουμε μία έκθεση που θα γίνει ομόφωνα δεκτή και αυτό είναι το επιστέγασμα των προσπαθειών μας να εξυπηρετήσουμε τους πολίτες. Και από τις συναντήσεις με τις αρχές. Είχαμε πολύ σε βάθος διαλόγους με τη τις γεωλογικές έρευνες σχετική αυτή η υπηρεσία στην Πολωνία, την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες περιφερειακές αρχές. Και επίσης ενημερωθήκαμε μόλις πριν από ένα τέταρτο από την Πολωνική Αποστολή ότι θα συμβάλλουν και με δύο ακόμα στοιχεία. Δηλαδή πρώτον με πρόσθετες πληροφορίες για τα, το εξορυκτικό πρόγραμμα και το σχιστολιθικό αέριο και κάτι που είναι ακόμα αρκετά νεφελώδες και αφορά μια συγκεκριμένη επιστολή που δεν θέλω τώρα να την πολύ συζητήσω. Τέλος, πριν μπούμε στο, στις λεπτομέρειες του περιεχομένου, πάντοτε τα δύο μέλη μας, συν τους άλλους διακεκριμένους συναδέλφους, όλοι ανέφεραν ότι εμείς πήγαμε στην Πολωνία όχι ως κριτές, δικαστές, ούτε ως εισαγγελείς πήγαμε για να δείξουμε την εκτίμησή μας σε ένα ε, εξέχον κράτος μέλος. Εγώ προσωπικά αισθάνομαι πολύ κοντά στην Πολωνία χάρη στην ιστορία μου και τις ιδιαίτερες σχέσεις της χώρας μου με την Πολωνία και επειδή η Πολωνία ε, χρησιμοποίησε τη χώρα μου στη Πολωνική εξορία ώστε να βρει καταφύγιο σε ε, μια εποχή όπου ταλαιπωρήθηκε η ελίτ της Πολωνίας και γι' αυτό είχαμε ε, συνομιλίες με απόλυτο σεβασμό προς όλους, χωρίς να υπάρχουν προκαταλήψεις, προκατασκευασμένες ιδέες πριν υπάρξει ε, ουσιαστικός διάλογος και με τους αναφέροντες και με τις αρχές. Σας καλώ όλους να διαβάσετε πολύ προσεκτικά την ουσία της έκθεσης, το περιεχόμενο, το οποίο νομίζω ότι λίγο θα τροποποιηθεί, το ελπίζω τουλάχιστον, λίγο μόνο. Σας καλώ να συμβάλλετε κι εσείς, να συμμετέχετε και να το εγκρίνετε, να εγκρίνετε την έκθεση όταν έρθει η ώρα με τρόπο επικοδομητικό και φιλικό για να αποδειχθεί ότι η Επιτροπή Αναφορών είναι ένας χώρος που εξυπηρετεί τα μελήματα των ε, πολιτών. Δύο λόγια μόνο τώρα για αυτό που φαίνεται να είναι ε, το, η πιο προβληματική πτυχή από την επισκεψή μας στην Πολωνία. Καταρχήν υπάρχει σαφής έλλειψη επικοινωνίας μεταξύ των αρχών και των πολιτών παύλα αναφερόντων. Και ένα παράδειγμα είναι ότι στην περιφέρεια της ε, Λέτια οργάνωσαν 12 δημοψηφίσματα. Η έκβαση από την συμμετοχή σε αυτά τα δημοψηφίσματα ήταν, η συμμετοχή δηλαδή 92 με 99% του πληθυσμού, που είναι ένα, α, α, διορθώνω, ήταν πάνω από το 60% οι συμμετασχόντες από όλο τον πληθυσμό και η αρνητική αντίδραση απόρριψης του έργου δηλαδή ήταν άνω του 60% σε όλα τα δημοψηφίσματα. Ήταν πάνω από το 60%. Έτσι λοιπόν το ρητορικό μου μάλλον ερώτημα είναι πώς να εμπιστευτούμε τη διαφάνεια και τη συμμετοχή των πολιτών και τις δημόσιες διαβουλεύσεις όταν είμαστε αντιμέτωποι με μια τέτοια πραγματικότητα. Και δεύτερον, και νομίζω και ο Chris Τέιλορ θα συμφωνήσει μαζί μου που είναι εδώ, ε, είναι ότι για το σχιστολιθικό, το σχιστολιθικό αέριο είναι κάτι που με μπερδεύει. Είναι σαν θρησκεία. Κανείς δεν έχει δικαίωμα να θέσει ερωτήματα για το σχιστολιθικό αέριο. Δηλαδή σαν να μην είναι θεμητό να τεθεί καμία ανησυχία, να διατυπωθεί κανένα πρόβλημα. Δηλαδή είναι λιγάκι μια θρησκευτική προσήλωση προς το σχιστολιθικό που δεν συνάδει με τους ενωσιακούς κανόνες που προβλέπουν διαφάνεια, διαβουλεύσεις ε, δημόσιες, ε, μελέτη επιπτώσεων περιβαλλοντικών, ε, εκτίμηση ΕΠΕ δηλαδή. Βεβαίως όλα, θα, θα συλλεγούν όλες οι πληροφορίες πριν επανέλθω και ευχαριστώ όλους όσοι ήρθαν σε αυτή την ωραία αποστολή στην ε, Πολωνία εκτός από ότι το Βρόσλαφ είναι μια όμορφη πόλη ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε λόγο να ξαναπάμε και στο Γκτάνσκ όχι όμως για να συναντήσουμε τους αναφέροντες πάντως έχουν μια αξιόλογη διοικητική ικανότητα, μια αξιόλογη ικανότητα να αφομοιώνουν τα ενωσιακά κονδύλια με έξυπνο τρόπο. Πρόκειται για μια πόλη πλήρως αποκαταστημένη, αναπλασμένη, με ωραίο αεροδρόμιο, στάδιο κλπ. κλπ. Είναι ένας χώρος που αγάπησα και τον αγαπώ. Γι' αυτό λοιπόν καλό είναι να δούμε την ουσία της επίσκεψης με ανοιχτό πνεύμα, ανοιχτή καρδιά και να καταλήξουμε σε συμπεράσματα όταν όλες οι συμβολές, συνεισφορές θα είναι επιτάπητος. Ευχαριστώ, Τζίνγκουε Μπάρτζοκ και ε, ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν προβλήματα με την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Καμιά φορά φαίνεται ότι η Επιτροπή μας ε, επιτυγχάνει ψηλούς στόχους. Χωρίς μικρόφωνο, κύριος Μποστινάρου. Χωρίς μικρόφωνο συνεχίζει ο κύριος Μποστινάρου. Πάντως ήταν μια μέρα τυχερή για μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Τέιλορ. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Μποστινάρου το προσωπικό και όσους συμμετείχαν στη διοργάνωση αυτής της εξαιρετικής ε, διερευνητικής αποστολής. Ο κ. Μποστινάρου ήταν πολύ ικανός και επιδέξιος ε, κεφαλής αυτής της αντιπροσωπείας. Και πριν ακόμα πάμε, με ενδιαφερόμουν πολύ για το θέμα. Το ταξίδι αυτό ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Μάλιστα έμεινα και μερικές μέρες παραπάνω εκεί και πήγα και στο Γκτάνσκ, στην περιοχή του Γκτάνσκ όπου συναντήθηκα με διάφορους ενδιαφερόμενους ακτιβιστές κλπ. Φαντάζομαι ότι όλοι πήρατε το blog μου, είδατε το blog μου, βρίσκεται στη, σελίδα μου στο ίντερνετ. Ε, έκανα και κάποιες ερωτήσεις εκεί. Ε, σας έχω στείλει τη διεύθυνση για το πρώτο τμήμα και το δεύτερο τμήμα. Το ένα τμήμα αφορά τα ορχεία και το άλλο τμήμα αφορά το σχιστολιθικό αέριο. Ε, η έκθεση είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στο Στρασβούργο αυτό το Σαββατοκύριακο στην Αυστρία και δεν είχα χρόνο να την διαβάσω έτσι λεπτομερώς σε βάθος. Οπότε θα περιοριστώ σε μερικά γενικά σχόλια προς το παρόν. Χωρίς συγκεκριμένη σειρά. Ίσως ε, θα έπρεπε να αναφερθούμε στις προτάσεις κομισιών που αναμένονται για την εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου. Αναμένονται για το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο περίπου. Δεκέμβρη λέει ο κ. Μποστινάρου, μάλιστα. Ίσως επίσης θα πρέπει να αναφερθούμε και στις αναθεωρήσεις ε, των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. κάτι δεν έγινε σωστά στην Πολωνία. Ο Βίκτορ είπε ότι σαν να πρόκειται για δογματική άποψη ε, αυτή που είναι υπέρ του, του σχιστολιθικού αερίου ε, πράγματι συμφωνώ απόλυτα είναι σαν ένα θέμα πίστης που δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει με επιστημονικά ή αντικειμενικά δεδομένα οπότε η δική μου αρχική ερώτηση ήταν αν είναι τόσο καλή αυτή η μέθοδος, γιατί δεν τη συζητάμε, γιατί αρνείστε να τη συζητήσετε. Γιατί αρνείστε να συζητήσετε τη ρηγμάτωση. Επίσης, χρειάζεται μια διευκρίνηση για τις μακροχρόνιες ε, ευθύνες ε, των ε, εγκαταστάσεων. Σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία, η ευθύνη ε, των εταιριών που κάνουν την εξαγωγή του αερίου είναι πολύ περιορισμένη χρονικά ενώ <laughs> οι ενδεχόμενες ε, συνέπειες είναι μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες. Ε, οι ευθύνες θα έχουν περάσει το κράτος πολύ νωρίς και θα πρέπει το κράτος να αναλάβει την επιδιόρθωση, την ε, επισκευή κλπ. Ε, τώρα, το θέμα της διαφάνειας. Τέσσερις μόλις ε, εβδομάδες δόθηκαν στο κοινό και στην κοινωνία για να γίνει διαβούλευση. Το δέχτηκαν αυτό, το παραδέχτηκαν και οι ίδιοι οι θύνοντες. Τέσσερις εβδομάδες για μια ολόκληρη χώρα είναι πραγματικά πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και ίσως θα έπρεπε να αυξηθεί. στις συστάσεις θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της σωστής διαβούλευσης και τη σημασία συμμετοχής της κοινωνίας. Στο, όπως, όπως ε, υπόθηκε, έγινε δημοψήφισμα στη Σιλεσία μεταξύ των 50.000 κατοίκων που πλήττονται περισσότερο και αυτό είναι σημαντικό. Και το δημοψήφισμα τι έδωσε, 95% ε, του, των ψηφοφόρων ήταν εναντίον του project, κάτι που είναι εντυπωσιακό, διότι το project αυτό θα ο δημιουργούς θα δημιουργούσε... Ε, δεν είναι εκπληκτικό μάλλον, γιατί το project αυτό θα καταργούσε τα πάντα. Θα κατέστρεφε ξενοδοχεία, δρόμου, ε, σχολεία, νοσοκομεία, γιατί θα δημιουργούσε τρύπε 200 μέτρων. Τώρα το ερώτημα είναι το υπόλοιπο 5% τι θεωρούσε ότι είναι καλό το project. τέλο πάντων, ε, γνωρίζουμε ότι εκεί υπάρχουν, υπάρχει και, ευρωπα, και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, δίδεται και ευρωπαϊκή χρηματοδότηση και θα πρέπει να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Τώρα, σε ό,τι φορά τις ειδικέ συστάσεις για το σχιστολιθικό αέριο. Με εντυπωσιάζει η ασυνέπεια της πολωνικής ενεργειακής στρατηγικής. Δεν ακολουθεί τις ε, ορθές ε, πρακτικές ε, που απαιτεί η ατζέντα του 2020 για τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Επιπλέον, έχασα το χαρτάκι μου. Η μείωση του διοξιδίου του άνθρακα αναφέρεται ε, στη στρατηγική μάλλον ακροθυγός. Νομίζω ότι θα χρειαζόταν να διευκρινιστεί περισσότερο. Θυμάμαι ότι στην παρουσίαση που έγινε εδώ στην Επιτροπή μας για την εξαγωγή σχιστολιτικού αερίου, ε, το κέντρο Tyndall στο Βόρεια Αγγλία μας είχε δώσει κάποια ε, δεδομένα αδιαμφισβήτητα και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο πλευράς κλιματικής αλλαγής το πιο ασφαλές σημείο για το σχιστολιθικό αέριο είναι να μείνει εκεί που είναι. Η εξαγωγή του, η εξόριξή του, ε, πλήττει τις προσπάθειες μείωσης διοξιδίου του άνθρακα. Αυτά τα πορίσματα δεν έχουν ληφθεί έπαρκος υπόψη. Θα ήθελα τα συμπεράσματα του Ερευνητικού Κέντρου Τίντλ να ληφθούν περισσότερο υπόψη στην Πολωνία. Αν θα ε, περιμένουμε κάποια πρόσθετα σχόλια από τις πολωνικές αρχές όπως είπατε και εγώ θα κάνω κάποια πρόσθετα σχόλια τις επόμενες εβδομάδες. Νομίζω όμως ότι η αποστολή αυτή ήταν πολύ καλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Τέιλορ. Ποιος άλλος θέλει να πάρει το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μετά από όλα όσα ακούσαμε από τις θαυμάσεις αυτές παρουσιάσεις, τι να προσθέσω. Είμαι ευγνώμη προς τον κύριο Μποστινάρου για τα σχόλιά του και τη συνεισφορά του στην αποστολή. Δεν το διάβασα ακόμα το έγγραφο. Από την παρουσίασή σας όμως ε, είδα ότι φτάσατε σε κάποια αποτελέσματα, σε κάποια συμπεράσματα. Και τελικά θα αντιμετωπιστούν πιστεύω οι ανησυχίες που και εσείς και ο κύριος Τέιλορ ε, παρουσιάσατε σήμερα. Ε, περιμένουμε πανημοπονησία να δούμε τα συμπεράσματα της συζήτησης σε κάνα δύο εβδομάδες. Με προκαλέσατε με θετικό τρόπο κύριε Τέιλορ. Γι' αυτό θέλω να προσθέσω λίγα ακόμα στοιχεία που περιγράφουν και το περιβάλλον στο οποίο βρεθήκαμε στην Πολωνία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πρωθυπουργό και ο Υπουργό Περιβάλλοντος, ο κ. Τούσκ δηλαδή, και ο Υπουργό ε, Περιβάλλοντος είχαν μία διαμάχη. Ο Πρωθυπουργό πιέζει τον Υπουργό να τροποποιήσει την νομοθεσία, ούτω ώστε να είναι πολύ πιο φιλική για τους επενδυτές ε, φυσικού αερίου με πολύ σκληρό τρόπο. το εσύ του λέει, γιατί αλλιώς θα, θα φέρω κάποιον άλλο να το κάνει. Επίσης υπάρχει ένα σχέδιο τροπολογίας όπου οι μη κυβερνητικέ οργανώσεις λέγεται ότι μπορούν να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση αν λειτουργούν πάνω από ένα χρόνο. Άρα δηλαδή υπάρχει περιορισμός στη συμμετοχή των μη κυβερνητικών οργανώσεων να συμμετάσχουν στη δημόσια αυτή διαβούλευση, συζήτηση και αυτό είναι ανησυχητικό κατά τη γνώμη μου. Αυτό είναι το δεύτερο. Τρίτον, όταν ήρθαμε με, σε επαφή με τους γεωλόγους της Πολωνίας, ενημερωθήκαμε μόνο για κάποια στοιχεία για την εξόριξη και την διερεύνηση. Αλλά ούτε μία λέξη δεν μας είπαν για τη φάση της εκμετάλλευσης στην οποία βρισκόμαστε που είναι η πιο προβληματική, ε, που δημιουργεί και τα περισσότερα προβλήματα στο περιβάλλον. Ακόμα πιο ανησυχητικό, μας είπαν οι εκπρόσωποι του Πολωνικού Γεωλογικού Ινστιτούτου ότι η τεχνολογία και η τεχνική που θα χρησιμοποιηθεί τελικά στην Πολωνία είναι πιο προηγμένη από αυτή που χρησιμοποιήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Την περασμένη εβδομάδα η κυρία Ράσελ, εκπρόσωπος της Ευρών, με ρώτησε κάποια πράγματα. Ε, μου είπε ότι είναι επενδυτής, ενδιαφέρεται για αυτό το project στην Πολωνία. Εγώ δεν το ήξερα, αλλά η Σεβρών μας είπε ότι ναι, συμμετέχει σε αυτό το πρόγραμμα. Το Γεωλογικό Ινστιτούτο της ε, Πολωνίας μας είπε λοιπόν ότι υπάρχουν ε, στη διάθεση της Πολωνίας πιο προηγμένες τεχνολογίες από αυτές που χρησιμοποιούν σήμερα οι Αμερικάνοι. Και κάτι καλό. Είχα μια συνάντηση σε ένα χωριό, όχι για να μιλήσουμε για την ευημερία, και το υψηλό επίπεδο, υψηλό βιωτικό επίπεδο στην περιοχή, αλλά ήρθαμε σε επαφή με 100 κατοίκους από όλη την περιοχή. 127 ε, για την ακρίβεια ήταν συμμετέχοντες. Τηλεοπτικά κανάλια, τεράστια κάλυψη από τον τύπο της περιοχής κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μας. Όλα τα σχόλια ήταν θετικά που ακούστηκαν. Αυτό σημαίνει ότι για τη συμμετοχή μας εννοώ, για την προσπάθειά μας. Άρα αυτό δείχνει ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από το ενδιαφέρον μας, το πραγματικό ενδιαφέρον, όχι προπαγάνδα και ιδεολογήματα. Επίσης, οι εκπρόσωποι του Πολωνικού Γεωλογικού Ινστιτούτου μας είπε ότι η πολωνική κυβέρνηση είναι αντίθετη σε κάθε τροπολογία στην περιβαλλοντική μελέτη αντικτύπου που, που μιλάει για τα προβλήματα του σχιστολιθικού αερίου και δεν θέλει να υιοθετήσει νέα νομοθεσία για το σχιστολιθικό αέριο. Όλα αυτά μαζί τι μας λένε. Η εικόνα είναι λίγο πιο ανησυχητική από ότι όταν τα βλέπουμε όλα αυτά τα στοιχεία χωριστά. Λέω να σταματήσω εδώ. Ευχαριστώ τον κύριο Βαουέσα ακόμα μια φορά. Γιατί δείχνει ευήκονους για τα προβλήματα και τις ανησυχίες των Ευρωπαίων πολιτών. Καλό παράδειγμα αυτό θα είναι για τις, υπόλοιπες, για τις επόμενες αποστολές που θα έχουμε. Θα βάλω λοιπόν το σημείο αυτό στην επόμενη συνεδρίασή μας και σήμερα σταματάμε εδώ τη συζήτηση. Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι τα τρία σημεία για τις αναφορές που αναφέρονται στο σημείο 5 και 6. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την ίδια καταγγελία. Στο σημείο 5 έχουμε μία αναφορά ε, που που υποβάλλεται από την Ένωση Ριφιουτάρση. Δεν είναι παρόντες συντάκτες ε, για αυτή την αναφορά, αλλά είναι παρόντες οι συντάκτες της αναφοράς 6. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο στους παρευρισκόμενους της ε, αναφοράς 6 για 5 λεπτά ε, στους δύο αυτούς λοιπόν κυρίους για να μας μιλήσουν για το θέμα τους. Κυρίες και κύριοι. Είμαι ιερέα στην Καθολική Εκκλησία στην επαρχία της Νάπολης, στην περιοχή Καϊβάνο, που είναι ένα χωριό που έγινε διαβόητο δυστυχώς, γιατί σε, αυτή, σε αυτό το χωριό, όπως και σε όλη την επαρχία της Νάπολης, στη Βόρεια Νάπολη, στην Καζέρτα, ζούμε ένα ανθρωπιστικό δράμα εδώ και χρόνια, που δυστυχώς το αποσιωπούν οι πάντες. Τα τελευταία χρόνια, μετά από μία εκστρατεία της εφημερίδας Αβενίρε, αυτό το πρόβλημα αρχίζουμε να το συζητάμε λίγο παραπάνω, γιατί συζητήθηκε μέσω της εφημερίδας. Η περιοχή μας επί χρόνια μαστίζεται από την Καμόρα. Έχουμε άτιμους βιομηχάνους, έχουμε συνενοχή διεφθαρμένων πολιτικών ή αμαθών πολιτικών Όλα αυτά λοιπόν επέτρεψαν στις, στα χωριά μας, στην επαρχία μας που ήταν τόσο πλούσια, τόσο όμορφη, να θαυτούν χιλιάδες τόνων απορρίμματα βιομηχανικής φύσεως που είναι πάρα πολύ τοξικά. Θαύτηκαν λοιπόν, κυριολεκτικά, και το αποτέλεσμα είναι ότι αναδύονται τοξικοί καπνοί Σας φαίνεται περίεργο και είναι πραγματικά περίεργο. Εμείς, όποιοι οι απλοί άνθρωποι, οι ιερείς, οι γιατροί, οι οικογενειακοί γιατροί, συνειδητοποίησαμε ότι τα τελευταία χρόνια η θνησιμότητα λόγω καρκίνου, λόγω όγκων αυξήθηκε εκθετικά. Αρρωσταίνουν τα παιδιά, αρρωσταίνουν οι νέες γυναίκες, οι νέες μαμάδες και μεταφέρουμε στο νεκροταφείο χιλιάδες άτομα πριν από τη φυσιολογική του ώρα. Ο, ο κόσμος έρχεται κλαίγοντας σε εμά. Γιατί πια, και το λέω με θλίψη, γιατί δεν έχει καμία εμπιστοσύνη σε τίποτα και σε κανένα. Δυστυχώς, η φωνή μας είναι μία δύναμη φωνή. Και φτάσαμε εδώ και σας το λέω πραγματικά από καρδιάς. Με την δύναμη της απελπισίας. Όταν η κυρία Ματσόνη έφτασε στην εκκλησία μου πέρυσι, σκεφτήκαμε εκεί με τους συγχωριανούς ότι η Ευρώπη έρχεται να μας βοηθήσει. Η καμπάνια δεν έχει πια πέντε επαρχίες, έχει έξι. Η έκτη είναι η γη των καπνών, των αναθυμιάσεων και των δηλητηρίων. Είναι η γη μου. Η γη αυτή που δεν μας είχε ποτέ προδώσει, ξαφνικά έγινε εχθρός μας. Η δασοκομική υπηρεσία αυτές τις μέρες ε, βρήκε, βρήκε σε καλλιεργήσιμους αγρούς ε, που καλλιεργούνται ντομάτες και σπαράγγια. Σκεφτείτε ότι αυτά εξάγονται στην Ευρώπη, έτσι. Τα έλεγξε αυτά τα προϊόντα και βρήκαμε ότι είναι δηλητηριώδη. Χθες, Κυριακή, Εγώ φωτογράφησα τις ε, ντομάτες αυτές και τις έστειλα σε εφημερίδες. Αυτές οι... Αυτή η κατάσταση που συμβαίνει πια σε εμά δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι περίπτω να πούμε ότι άμεσα υπεύθυνοι είναι οι δήμοι, οι κοινότητε, οι, οι δήμαρχοι, οι οποίοι έχουν στήσει την άσπρη σημαία, που έχουν παραδοθεί λέγοντας ότι δεν έχουν πια τη δύναμη να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Το περασμένο μήνα βρέθηκαν 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα τοξικών απορριμμάτων βιομηχανικής φύσεως θαμμένα. Μιλάμε ε, για απόβλητα που παράγονται στις βιομηχανίες μας του Βορρά και φτάνουν σε μας και που ε, βιομηχανίες και επιχειρήσεις που ζουν μέσα σε ένα καθεστώς ε, φορολογικής ε, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Αυτό το δηλητηριώδες, αυτή τη δηλητηριώδη ανάσα τη ζούμε, την αισθανόμαστε πάνω στο σβέρκο μας. Σας παρακαλούμε να λάβετε υπόψη αυτή την έκκληση, Πρόεδρε. Είμαστε και εμείς Ευρωπαίοι, Πρόεδρε, και σε αυτή την περιοχή δεν μπορούμε να ζήσουμε πια. Έχουμε δημιουργήσει εκατοντάδες επιτροπές. Η Καθολική Εκκλησία ασχολείται και γίνεται ας πούμε ο εκπρόσωπος αυτών των απελπισμένων φωνών. Ο επίσκοπος με τον αρχιεπίσκοπο της Νάπολης ε, υπέγραψαν ένα πολύ σκληρό έγγραφο λέγοντας ότι ανησυχούν πραγματικά για όλα όσα συμβαίνουν. Φτάσαμε εδώ, φτάσαμε σήμερα το πρωί και θα φτάσουμε σήμερα το βράδυ στην, στο χωριό μας. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φτάσω μέσα σε μια, μια μέρα στις Βρυξέλλες για να κάτσω μια μέρα και να φύγω το βράδυ μόνο. Σας μίλησα για αυτές τις επιτροπές. Και εγώ ως κληρικός Είμαι λίγο ο πνευματικός σε αυτές τις συγκεντρώσεις. Ασχολούμαι με τα άτομα τα οποία δεν αντέχουν άλλο. Νέους χωρίς ελπίδα, ανθρώπους που έχουν απελπιστεί. Ε, σας ζητώ όσο υπάρχει χρόνος να κάνετε κάτι. Ο κύριος που μίλησε προηγουμένως είπε κάτι πολύ όμορφο. Το είχα σκεφτεί κι εγώ σε αυτά τα γυάλινα μέγαρα όπου λαμβάνονται αποφάσεις πρέπει κάποια στιγμή ο κόσμος να συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να μειώσει τις αποστάσεις ανάμεσα σε αυτά τα γυάλινα παλάτια και στον πραγματικό και απλό λαό. Πρέπει να σταθείτε δίπλα σε αυτό τον κόσμο. Η Νότια Καζέρτα και η Βόρεια Νάπολη έχουν γίνει περιοχές δηλητηριασμένες. Φοβόμαστε ακόμα να βγούμε για να ψωνίσουμε. Δεν ξέρουμε καν ποιες είναι οι περιοχές οι αγροί, οι δηλητηριασμένοι. Πρέπει να ξέρουμε ποια είναι τα μέρη, οι... τα χωράφια, τα οποία δεν είναι δηλητηριασμένα, τόσο ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να καλλιεργήσουν εκεί. Να κάνουμε... Ε, να βελτιώσουμε τα εδάφη μας ε, η βελτίωση αυτή δεν γίνεται. Τα λεφτά εξαφανίζονται. Πρέπει να μπλοκαριστεί η μεταφορά αυτή βιομηχανικών τοξικών αποβλήτων από το βορρά στις δικές μας επαρχίες. Όποιος έκανε λάθος επίσης πρέπει να πληρώσει. Είναι ανυπόφορη αυτή η κατάσταση. Είναι ανυπόφορο να λέμε ότι ναι έκανες λάθος αλλά πήγαινε σπίτι σου, δεν πειράζει. Ο λαός της Νάπολης και της Καζέρτα στην καμπάνια σας κάνει αυτή την έκκληση και σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Ευχαριστώ, εδεσιμότατε Μαουρίτσιο. Ο κύριος Μαρφέλα για πέντε λεπτά. Σας ευχαριστώ πρόεδρε, σας ευχαριστώ που με ακούτε, που μας ακούτε. Ως τεχνικός ε, απόκειται σε μένα να εξηγήσω αυτά που είπε ο εδεσιμότατος Μαουρίτσιο. Κάνω έκκληση σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτως ώστε να ασχοληθεί με την δέουσα προσοχή ε, με αυτό το θέμα. Δεν μιλάμε για αστικά απόβλητα, για τα οποία όλοι ανησυχούμε, αλλά να δώσετε τη μέγιστη δυνατή προσοχή στην Ευρώπη, στην παραγωγή και στη σωστή διάθεση βιομηχανικών αποβλήτων, έτσι, όχι αστικών, που παράγονται στην Ευρώπη και στην Ιταλία φτάνουν πλέον 140 εκατομμύρια τόνοι αποβλήτων σε σχέση με τα 30 εκατομμύρια τόνων αστικών αποβλήτων. Και για αυτά τα 140 εκατομμύρια ανησυχούμε. Νομίζω ότι είμαστε οι ντροπιασμένοι όλου του κόσμου, γιατί δεν διαθέτουμε σωστά τα απορρίμματα. Εδώ και 30 χρόνια και πλέον η καμπάνια, η χώρα, το λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού μαζί με την Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια έχει γίνει η βιομηχανική χωματερή αυτών των αποβλήτων. Μιλάμε για απόβλητα που παράγονται σε καθεστώς φορολογικής αποφυγής. Εμείς παράγουμε στην Ιταλία 138 τόνους βιομηχανικών αποβλήτων. Κυκλοφορούν ελεύθερα ως εμπορεύματα αυτά τα απόβλητα. Σας παρακαλώ, αγαπητοί ευρωβουλευτέ, προσοχή σε αυτό το θέμα. Εάν λάβουμε υπόψη μα ότι η φοροδιαφυγή στη χώρα μας είναι πολύ υψηλή, είναι το περίπου το 30% κατά μέσο όρο. Αυτό το γεγονός ε, μας επιβάλλει να λάβουμε υπόψη μας τι γίνεται με τα 30-35 35 τονους αποβλήτων το χρόνο, εκατομμύρια τόνους το χρόνο που δεν ε, διαθέτονται σωστά. Από τις πιο αρχές περιοχές είναι η καμπάνια. Ε, λίκνο του πολιτισμού, η πατρίδα του Οράτιου και του Πομπίου και της ε, Πομπίας. Ε, ε, εκεί βρίσκεται η πόλη της Πομπίας. Μην τα ξεχάσετε αυτά. Πριν από ένα χρόνο Αποδείξαμε ότι οι 11 πολεμιστές που σκοτώθηκαν μπλοκάροντας τα στρατεύματα του Ανίβα, ε, αυτή η τάφη αυτών των πολεμιστών ε, είναι δηλητηριασμένη από διοξίνη. Αυτή είναι η πατρίδα των πολεμιστών. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες νίκες του αρχαίου κόσμου απέναντι στον Ανίβα. Δεν μπορούμε να διαθέσουμε σωστά όπως πρέπει τα απόβλητα. Ε, το αποτέλεσμα είναι τοξική καπνή και θυμιάσει. Σας παρουσιάσαμε μία σειρά από έγγραφα όπου παρουσιάζουμε τα γεγονότα και ζητάμε την ε, ε ταυτόχρονη παρέμβαση όλων των ε, αρμόδιων Υπουργείων της Ιταλίας. Αλλά επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει τη δέουσα προσοχή στο πρόβλημα της καμπάνιας. Γιατί αν δεν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι δεν διαθέτονται σωστά τα βιομηχανικά απόβλητα της Ευρώπης. Και αν δεν εντοπίσουμε σωστά την πηγή και το πρόβλημα, δεν μπορούμε ποτέ να διορθώσουμε. Να το διορθώσουμε. διαπιστώσαμε ότι επί 30 χρόνια υπάρχει αυτό το πρόβλημα και δεν το διορθώνουμε. Αυτό είναι έλλειψη πολιτισμού. Δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις. Δεν έχουμε σωστές εγκαταστάσεις για τα αστικά απόβλητα. Αλλά επιπλέον στην καμπάνια υπάρχουν α, πολλά προβλήματα με τις εγκαταστάσεις όπου διαθήκενται τα βιομηχανικά απόβλητα. Παραδείγματο χάρη του αμίαντου. Σε μια εγκατάσταση εκεί διαθέτουμε τον αμίαντο. Προσπαθούμε από, τους, όλο το τροχαίο υλικό της ε, Ιταλίας να αφαιρέσουμε τον αμίαντο και να τον στείλουμε σε αυτή την εγκατάσταση στην περιοχή μας. Οι εκκλήσεις μου είναι οι εξής. Προσοχή. Πρέπει να γίνεται σωστή διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων και σωστή χνηλασιμότητα να υπάρχει των αποβλήτων αυτών στην Ευρώπη. Γιατί όταν υπάρχει χνηλασιμότητα δεν ξέρουμε από πού προέρχονται τα προβλήματα και πού είναι η πηγή και πώς κυκλοφορούν οι ροές. Δεύτερον, προσοχή. Πρέπει να ασχοληθούμε με τη σωστή διάθεση των αστικών αποβλήτων, φυσικά, αλλά Μην ξεχνάτε ότι η παραγωγή βιομηχανικών αποβλήτων σε σχέση με τον αστικό είναι 4 προς 1. Επομένως πρέπει να προσέξουμε κυρίως την σωστή διάθεση των βιομηχανικών αποβλήτων. Επίσης, με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία που έχουμε στην περιοχή μας, φαίνεται ότι ο πληθυσμός δηλητηριάζεται πια. Είναι μία περιοχή η οποία πλήττεται από την μεταφορά τέτοιων αποβλήτων και τη διάθεση τέτοιων αποβλήτων. Σας παρακαλούμε και τις περιφερειακές αρχές μας αλλά και τις τοπικές αρχές μας να ασχοληθείτε, να δώσετε σημασία στις ε, επιδημιολογικές αυτές μελέτες. Πρέπει να γίνει μια ακόμα ευρύτερη επιδημιολογική μελέτη. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η καταστροφή στην ε, περιοχή μου δεν έχουμε σοβαρά επιδημιολογικά στοιχεία για την καμπάνια. Ούτως ώστε να υπάρξει και η σωστή πολιτική και να βρουν οι πολίτες πάλι την ελπίδα τους. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε και σας οικετεύω να δώσετε τη μεγαλύτερη προσοχή στο θέμα της ελεύθερης κυκλοφορίας βιομηχανικών αποβλήτων. Κυκλοφορούσαν εμπορεύματα αυτά. Προσοχή, γιατί και στην Ευρώπη δεν υπάρχει νομοθεσία για περιβαλλοντικά δικήματα. και δεν έχουμε παρκώς αυστηρές κυρώσεις. Μπορούμε κάλλιστα λοιπόν να, διολο... να δηλητηριάζουμε ολόκληρους πληθυσμούς στην Ευρώπη Μπορούμε να ασχολούμαστε πολύ ας πούμε τον εντοπισμό των ναρκωτικών, αλλά δεν ασχολούμαστε καθόλου με το πρόβλημα αυτό το περιβαλλοντικό λόγω των βιομηχανικών αποβλήτων. Είναι ο δεύτερος λόγο θανάτων ε, λόγω περιβαλλοντικών αδικημάτων. Ο κύριος Μαγκανάρο από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε το θέμα των βιομηχανικών αποβλήτων στην καμπάνια. Έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση, είναι ακόμα ανοιχτή αυτή. Στις 20 Ιουνίου η Κομισιόν αποφάσισε να παραπέμψει την Ιταλία για δεύτερη φορά ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Με βάση τις πληροφορίες που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ξεκινάμε από τις πληροφορίες που μας έδωσαν οι ίδιες Ιταλικές αρχές, προκύπτει ότι δεν έχουν λυθεί ακόμα τα κατάλληλα μέτρα, ούτως ώστε να εξασφαλίσουμε ότι μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα η Ιταλία θα μπορέσει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του 2010. Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο ερώτημα τώρα της παράνομης διάθεσης των ε, αποβλήτων και κυρίως βιομηχανικών αποβλήτων στην καμπάνια, κυρίως σε ό,τι αφορά αυτό το πρόβλημα των καπνών και αναθυμιάσεων, η Κομισιόν με βάση τις ε, συνεχείς επαφές που έχει με τις ταγικές αρχές για αυτό το θέμα και το πρόβλημα της καμπάνιας, ζήτησε διευκρινήσεις και έκανε έκκληση και παρότρινε τις εθνικές αρχές να κάνουν το καταδύναμη, τόσο ώστε να ληφθούν τα μέτρα για να εξασφαλίσουμε μια μόνιμη παρακολούθηση της καμπάνιας, ούτως ώστε να προβλέψουμε και να σταματήσουμε την παράνομη αποτέφρωση, την παράνομη ταφή επίσης των αποβλήτων αυτών. Με βάση τις πληροφορίες που μας έδωσαν οι Ιταλικές αρχές, τον Οκτώβριο του 2012 δημιουργήθηκε ένα συντονιστικό μηχανισμός στην καμπάνια με τις ε, τοπικές αρχές και με... εμπλέκεται και η κεντρική κυβέρνηση καθώς και οι οργανώσεις, ούτως ώστε να υπάρχουν περιπολίες πιο τακτικές πιο συστηματικές, πιο πλαισιωμένες ε, σε ολόκληρη την καμπάνια. Από ό,τι φαίνεται αυτές οι περιπολίες σταμάτησαν, έγιναν διάφορες καταγγελίες γιατί υπήρξαν απαγωγές. Δηλαδή ε, εξαφανίζονται ε, εξαφανίζονται ολόκληρα φορτία αποβλήτων στην Νάπολη και στην Καζέρτα. Σε ό,τι αφορά τη σωστή διαχείριση των βιομηχανικών αποβλήτων στην καμπάνια, η Κομισιόν πίεσε επίσης τις τοπικές αρχές για να δημιουργήσουν και ένα ε, ειδικό σχέδιο διαχείρισης. Η καμπάνια τον Ιανουάριο του 2012 υιοθέτησε ένα σχέδιο για τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, αλλά παρουσίασε στην ε, Κομισιόν επίσης και ένα προσχέδιο για την ε, διαχείριση των ειδικών αποβλήτων. Πρόσφατα η Κομισιόν ζήτησε από τις Ιταλικές Αρχές να ενημερωθεί για τις ε, διαπραγματεύσεις ε, που πρέπει να γίνουν για να υιοθετηθεί αυτό το σχέδιο. Γιατί ενώ το σχέδιο για τα αστικά απόβλητα υιοθετήθηκε, όπως σας είπα, τον Ιανουάριο του 2012, το σχέδιο για τα ειδικά απόβλητα για την καμπάνια δεν έχει ακόμα υιοθετηθεί και η Κομισιόν ζήτησε από τις Ιταλικές Αρχές να την ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν για την κατάληξη αυτού του σχεδίου για τα ειδικά απόβλητα. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Όκεν. Ευχαριστώ. Ε. Δανέζικα uh, uh, θα μιλήσω. Καταρχήν να ευχαριστήσω τους αναφέροντες που ήρθαν στην Επιτροπή μας η υπόθεση είναι παλιά. Αυτά τα τερατώδη τα ακούμε εδώ και χρόνια. Και όταν πήγαμε σε αποστολή στην Νάπολη, δεν θυμάμαι πόσος καιρός είναι και συναντήσαμε τότε αναφέροντες εκεί. Ήταν μια σύντομης διάρκειας αποστολή, αλλά ενημερωθήκαμε ε, κατά μια μακρά πρωινή συνεδρίαση όπου ήρθαν και παρουσίασαν τις καταγγελίες τους οι αναφέροντες και καταλάβαμε στο τέλος ε, της συνάντησης ότι εδώ είναι τεράστια τα προβλήματα. Και στην ίδια την πόλη της ε, Νάπολης είχαν αναλυθεί πρωτοβουλίες για συλλογή από πόρτα σε πόρτα. Επίσης υπήρχε ένα σύστημα συλλογίστων των αποβλήτων όπου δεν καίγονταν όλα, αλλά έκανε ένα διαχωρισμό των ε, διαφόρων κατηγοριών αποβλήτων ε, από την πόλη και κάποια απόβλητα τα παραλάμβαναν οι γειτονικέ πόλεις. Αλλά και εδώ είναι το πιο ε, τρομερό και αρνητικό που είδαμε στην αποστολή. Φαίνεται ότι είναι αδύνατον να βρεθεί κάποιος υπεύθυνο για την κατάσταση αυτή. Στη Ρώμη ήρθε ο υπουργό και ρωτούσαμε ποιος είναι υπεύθυνο και τον μπαλάκι το άρπαζαν και το πέταγε ο ένας τον άλλον και όχι δεν φταίμε εμείς και είναι αρμόδιος ο δήμαρχος και υπεύθυνη ε, για αυτά τα θέματα στην Καμπανία και είπαν ότι 450 δήμαρχοι από την Καμπανία θα έπρεπε να ε, συνεννοηθούν για να αποφασίσουν. Για όνομα του Θεού, αν ισχύει αυτό, δεν θα λυθεί το πρόβλημα στην Ιταλία ποτέ. Αν δεν γίνει δηλαδή διοικητική μεταρρύθμιση στην Ιταλία, δεν θα μπορέσει να βρεθεί ο υπεύθυνο και να κατονομαστεί και δεν θα γίνει τίποτε, άρα το πρόβλημα παραμένει. Ίσως η Ιταλία να περηφανεύεται για το αποκεντρωμένο σύστημά της όπου ο καθένας είναι υπεύθυνο για τη δική του τη γονίτσα, αλλά βλέπουμε όμως και το αρνητικό της αποκέντρωσης. Εμείς παρακολουθήσαμε το θέμα εδώ και καιρό. Είδαμε τη ζημιά που έχει γίνει ε, λόγω της λανθασμένης, της πολύ λάθος αντιμετώπισης και την πρώτη φορά που πήγαμε και η Γιούντιθ Μέρκες και ο Πίτερ Γιάν και εγώ που πήγαμε την πρώτη φορά και μας είπαν τότε ότι πρόκειται για επικίνδυνα απόβλητα από τη Βόρεια Βιομηχανική Ιταλία και η μαφία κάνει τη διοικητική ε, διεκπαιρέωση και διακίνηση των τοξικών. Κάπου έπρεπε να πάνε και ίσως ε, τα ποντίζουν στη θάλασσα έξω από την Άπολη, παρόλο που είναι επικίνδυνα τα απόβλητα και κάποια τα καίνε. Όμως δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με αυτή την υποκριτική στάση και να επαναλαμβάνουμε το ίδιο μάντρα ότι πρόκειται για περιφερειακή αρμοδιότητα, ότι οι ΟΤΑ πρέπει να το λύσουν όταν είναι προφανές ότι υποφέρει ο κόσμος στην περιοχή λόγω αυτής της έλλειψης στην επεξεργασία των αποβλήτων. Ε, Υπάρχουν δυνατότητες και σε αυτή την περιφέρεια να λυθεί το πρόβλημα, όπως και σε άλλες περιφέρειες. Όταν μιλάμε για τον, με τον τόπιο πληθυσμό εκεί, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ καλή θέληση. Οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να αναλάβουν την ευθύνη για τα αποβλητά τους, αλλά στο βαθμό που όλα χάνονται μέσα σε αυτή την ομίχλη της ανευθυνότητας, δεν μπορεί να γίνουν πράγματα ακόμα και οι δήμαρχοι εκεί ε, δεν ε, έχουν αρμοδιότητα να ε, παρακολουθούν τους χώρους, τα φύση κλπ. Η Κομισιόν λέει ναι αρχίσαμε τη διαδικασία επί παραβάση λοιπά». Ή αυτά λέει το δικαστήριο και εμείς σκεφτήκαμε και εμείς θεωρούμε. Ε, αυτά είναι δηλώσεις που διαιωνίζονται χωρίς να συμβαίνει κάτι πρακτικό στο τοπικό επίπεδο εκεί που βρίσκεται το πρόβλημα. Νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε ότι υπάρχουν λόγοι πολύ συγκεκριμένοι για αυτή την κατάσταση και εκεί όπου έχει γίνει πρόοδος και όπως το, στην ίδια την πόλη της ε, Νάπολης ε, αποδεικνύεται ότι υπάρχουν λύσεις. Ελπίζω, γιατί ήταν τότε λίγο εύθραυστη λύση όταν είχαμε πάει εμείς, ελπίζω να εξακολουθεί να υφίσταται. Πάντως αυτές οι δομές πρέπει να ενισχυθούν. Ε, όμως είναι πάρα πολύ αποθαρρυντικό να καθόμαστε εδώ εμείς οι ευρωβουλευτές και ενώ επίσημα δεν έχουμε ευθύνη για την επεξεργασία των αποβλήτων στην Ιταλία, όμως παρόλα αυτά έχουμε ευθύνη όταν έρχονται σε εμά με τις καταγγελίες τους οι αναφέροντες. Και δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, όσο και αν είναι δραματικό αυτό. Αλλά πέρα από τα επικίνδυνα απόβλητα έχουμε και βουνά ολόκληρα οικολογικών όπως λέγονται αποβλήτων. Είναι βουνά στην περιοχή. και αν δεν καίγονται κατά από τις άθλιες συνθήκες που είδαμε, ε, τι γίνονται. Αλλά και με την καύση καταστρέφεται η θαυμάσια περιοχή της Καμπανίας. Ευχαριστώ κύριος Μποστινάρου. Yes, we can Ας αλλάξουμε τη σειρά. Ευχαριστώ Βίκτορ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η κατάσταση είναι απογοητευτική, αποθαρρυντική, εξοργιστική και η Κομισιόν βέβαια έκανε τη δουλειά της, ε, κίνησε διαδικασία επί παραβάση, αλλά θα πρέπει να ε, υπάρχουν δε και κονδύλια διαθέσιμα ε, για την περιοχή, για την αποκομιδή, επεξεργασία των αποβλήτων κλπ. Αλλά από την άλλη βλέπουμε ότι εδώ γίνονται διαδικασίες σε βάρος της περιφέρειας και του πληθυσμού. Εγώ όταν πήγα στην Άπολη είδα κάποιες ε, βελτιώσεις, είχαμε πάει με διερευνητική αποστολή για να δούμε το πρόβλημα ε, για τα οικιακά απόβλητα. Εκεί αναπτύχθηκε ένα σύστημα αποκομιδής ικανοποιητικό, αλλά με τα βιομηχανικά απόβλητα δεν είχε βρεθεί λύση τότε και από ό,τι καταλαβαίνω ούτε και τώρα έχει βρεθεί. Θα πρέπει λοιπόν να παραμείνουν οι αναφορές και θα πρέπει να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις στην τελική κυβέρνηση που είναι πολύ σημαντικές. Το είχα παρατηρήσει και τότε. Είχα ε, καταλάβει ότι τοξικά απόβλητα πήγαιναν στα νερά. Οι υπεύθυνοι της, ε, του χώρου απόθεσης έλεγαν ότι δεν ισχύει αυτό. Ε, τους ρωτήσαμε αν έγιναν δοκιμές για να δουν τι ισχύει και είπαν όχι δεν έγιναν δοκιμές. Ε, όπως είπε και ο χρειάζεται διαφάνεια σε αυτές τις υποθέσεις. Πρέπει να γνωρίζουμε που είναι μέσα στο έδαφος τα τοξικά απόβλητα. Πρέπει να το εξετάσουμε αυτό. Δεν μπορεί να λέμε ημέν ότι είναι εντάξει τα πράγματα, οι άλλοι να λένε όχι δεν είναι εντάξει. Θα πρέπει να γίνουν δοκιμές, να αποδειχθεί. Υπάρχουν πολλές επιστημονικές μέθοδοι για να διαπιστωθεί αν είναι ε, μολυσμένο το έδαφος. Ή είχαμε δει και ε, χωματερές με βουνά τα σκουπίδια. Και όταν τους ρωτήσαμε τι γίνεται με αυτά τα βουνά, δεν μου απάντησε, δεν μας απάντησε κανείς. Δηλαδή με την έννοια της διαχείρισης. Υπάρχουν λοιπόν τοξικά, ε, ε, είναι μολυσμένο ή υπάρχει μόλυνση τροφίμων, ε, υπάρχουν κάποια προβλήματα σε σχέση με νόσους που αυξάνονται σε ποσοστά στον πληθυσμό. Θα πρέπει κάποια στιγμή και η κεντρική κυβέρνηση να δει το θέμα και να διαθέσει και τα απαραίτητα κονδύλια. Επίσης θα πρέπει να παρακολουθούμε που πάνε τα βιομηχανικά απόβλητα και οι περιφέρειες και οι δήμαρχοι ε, φροντίζουν παρόλο που δεν μπορούν μόνο εκείνοι να λύσουν το πρόβλημα. Υπάρχουν ε, εγκληματικοί τοπικές οργανώσεις που παρεμβαίνουν και δημιουργούν πρόβλημα. Αν η χνευσιμότητα, η χνηλασιμότητα λοιπόν των, βιομηχών, των βιομηχανικών ε, αποβλήτων ε, και γιατί ε, υπάρχουν τώρα πια αναλύσεις και λένε ότι το 1 τρίτο, λένε οι αναλύσεις και οι έρευνες ότι το 1 τρίτο των βιομηχανικών αποβλήτων στην Ιταλία εξαφανίζεται. Πρέπει να υπάρχουν πιστοποιητικά. Πού είναι το 1 τρίτο. Και αυτές είναι οι σοβαρές εκτιμήσεις. Κανείς δεν ξέρει να πει πού πάνε αυτά τα απόβλητα. Πρώτον λοιπόν διαφάνεια, ίχνη λασιμότητα των βιομηχανικών αποβλήτων ε, Όποιος παράγει βιομηχανικά απόβλητα θα πρέπει να έχει πιστοποιητικό που θα αποδεικνύει πού πήγαν τα απόβλητά του. Πριν από δύο χρόνια δυστυχώς θα είχαμε πει τα ίδια αυτά. Ε, δεν ξέρω κυρία Πρόεδρε τι να κάνουμε, πρέπει να απευθυνθούμε στην κυβέρνηση, να καλέσουμε τον Υπουργό Περιβάλλοντος. Εγώ με τα δύο αυτά προβλήματα που ανέφερα διαπιστώνω ότι η ΟΤΑ και οι δήμαρχοι δεν μπορούν να λύσουν μόνοι τους το πρόβλημα. Ε, ήδη η Κομισιόν βέβαια έκανε τη δουλειά της αφού εκείνησε τη διαδικασία επί παραβάση, αλλά εκείνο που ενδιαφέρει είναι να αντιμετωπιστούν και οι εγκληματίες που βγάζουν χρήματα από τις παράνομες ε, και εγκληματικές τους δραστηριότητες. Αυτό είναι το αίτημα. Θα πρέπει λοιπόν να ασχοληθούμε, να δώσουμε συνέχεια στις δύο αναφορές, γιατί το είδαμε σε τελευταία ανάλυση όλοι είναι ε, εδική, ένας χώρος ιστορικός για την Ευρώπη και με αρχαία μνημεία ε, και δίπλα είναι τα σκουπίδια και τα επικίνδυνα απόβλητα. Ε, πρέπει λοιπόν να ξεπεράσουμε την αμηχανία που μας χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή και να έρθουμε σε επαφή με την κυβέρνηση για να καταπιαστούμε αυτό το σοβαρό θέμα. Ευχαριστώ κύριος Γιάρο, κύριος Μποστινάρου. Επιτρέψτε μου να μιλήσω στα ρουμανικά. Θα με καταλάβουν λίγο καλύτερα ενδεχομένως οι, Ιταλοί αναφέροντες. Αυτό που συζητάμε σήμερα αποδεικνύει καταδεικνύει μάλλον σαφώς το τι γίνεται όταν κατά συστηματικό τρόπο ένα κρατός μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραβιάζει όλη την κοινωτική νομοθεσία, τη σχετική κοινωτική νομοθεσία και την εθνική νομοθεσία. Ταυτόχρονα πρόκειται για μια συνεχή και επίμονη παράβαση της ε, κοινωτικής νομοθεσίας. Αυτό είναι το συμπέρασμα στο οποίο φτάνουμε τώρα. βλέπουμε να επανέρχεται στην ημερήσια διάταξή μας αυτό το θέμα της Ιταλίας. Έχουν αλλάξει τρεις κυβερνήσεις, Μπερλουσκόνη, Μόντι και η σημερινή κυβέρνηση. Κάτι που σημαίνει ότι συζητούμε εδώ και πολύ καιρό αυτή την πραγματικά προβληματική κατάσταση. Είναι σαφές ότι μόνο κατά παράβαση της κοινωτικής νομοθεσίας διατίθενται με αυτόν τον τρόπο τα βιομηχανικά απόβλητα. Κατά παράβαση όλων των σχετικών οδηγιών. Ακούμε με πολύ προσοχή το σκεπτικό των αναφερόντων. αλλά αναρωτιόμαστε πόσο καιρό ακόμα οι Ιταλικές αρχές θα συνεχίζουν να καταχρώνται της υπομονής μας. Και πόσο καιρό ακόμα η Κομισιόν θα συνεχίζει να καθυστερεί και να αναβάλει την απόφαση λήψης μέτρων, έστω και αυστηρών και σοβαρών μέτρων. Το πρόβλημα είναι πολύ σημαντικό και είναι το πρόβλημα της ανιχνευσιμότητας των αποβλήτων γενικότερα και των βιομηχανικών αποβλήτων ειδικότερα. Αυτό δεν αφορά μόνο την Ιταλία αλλά και τις υπόλοιπε χώρες. Και επηρεάζεται η διατροφική αλυσίδα αλλά και η υγεία μας και το περιβάλλον. Χρειάζεται να μπορούμε να ανιχνεύσουμε τα απόβλητα γενικότερα και τα βιομηχανικά απόβλητα ειδικότερα. Ένα τμήμα των βιομηχανικών αποβλήτων της Ιταλίας ξέρουμε πολύ καλά και ξέρω πολύ καλά ότι εξάγονται, εξάγεται στη χώρα μου, στη Ρουμανία. Η Ρουμανία όπως και η Ιταλία έχει ένα ισχυρό διοικητικό μηχανισμό αλλά η κατάσταση είναι ίδια. Υπάρχουν κανονισμοί, υπάρχουν οδηγίες, υπάρχει κοινοτική νομοθεσία και παρόλα αυτά εξακολουθούν με να είμαστε μάρτυρες τέτοιων καταστάσεων. Οπότε, πιστεύω ότι πρέπει αφενός να κρατήσουμε ανοιχτή την διαδικασία παραβάση. Δεύτερον, να καταστεί σαφές ότι η μαφία και το οργανωμένο έγκλημα εμπλέκονται άμεσα τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει θα πρέπει να τις ε, παραπέμψουμε, διαβιβάσουμε στην Επιτροπή ΚΡΙΜ που ασχολείται ακριβώς με το οργανωμένο έγκλημα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όχι μόνο με τη μαφία, γενικότερα με το οργανωμένο έγκλημα. Με αυτόν τον τρόπο ενδεχομένως θα μπορούσαν να εντοπιστούν οι αυτούργοι. Τέλος, Θα ήθελα και πάλι να παροτρύνουμε δραστήρια και ε, απροσχημάτιστα την Ιταλική κυβέρνηση να παρέμβει, να δώσει μια λύση. Είμαστε, συνδεόμαστε με ιστορικούς δεσμούς με την περιοχή αυτή. Δεν πρόκειται για την Αφρική ούτε για τις νέες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα συστατικό μέλος της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα μέλος όπου θεμελιώθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μην ξεχνάμε ότι πρόκειται για ένα πρόβλημα καθημερινότητας. Πρόκειται για ανθρώπους πραγματικούς, δεν βρίσκονται σε γυάλινους πύργους όπως εμείς. Θα πρέπει να τύχουν σεβασμού τα δικαιώματά τους και θα πρέπει να απαιτήσουμε μια απάντηση από τη νέα Ιταλική κυβέρνηση η οποία περηφανεύεται ότι αποτελεί πλειοψηφία των δύο μεγαλύτερων κομμάτων της χώρας. Συνεπώς, ας σταματήσουν να αλληλοκατηγορούνται ε, και να αποποιούνται των ευθυνών τους. Είναι ένα πρόβλημα μεγάλης εμβέλειας που ε, καθιστά την Ιταλία να ομοιάζει με αυτά τα αποτυχημένα κράτη τα οποία τα βλέπουμε από την αρχή της ιστορίας, από την εποχή του απογείου της Μεσοποταμίας μέχρι σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ πρόεδρε, θα μιλήσω τελικά. Όπως μας παρουσίασαν οι αναφέροντες, αλλά και οι ευρωβουλευτές, έχουμε συνεχή παραβίαση της νομοθεσίας. Αυτό είναι δεδομένο, είναι γεγονός, γίνεται εδώ και χρόνια, χωρίς καμία ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης. Πιστεύω ότι ένα από τα αίτια αυτής της κατάστασης οφείλεται στα σημερινά συστήματα ελέγχου, αλλά και στο σημερινό σύστημα που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την έναρξη διαδικασιών επιπαραβάση τις προθεσμίες, το χρόνο που χρειάζεται για να το κάνει, που είναι πάρα πολύ μεγάλος. Και επίσης ε, στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιεί μεθόδους αποτρεπτικές. Το σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό και δεν είναι προσαρμοσμένο στην κατάσταση που αντιμετωπίζουμε. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι παρά τις ε, τακτικές παρεμβάσεις της Επιτροπής και την επαφή που είχε με τις τοπικές αρχές, μέχρι στιγμής δεν είχαμε αυτά αποτελέσματα, σημαντικά αποτελέσματα. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, αυτά τα απόβλητα συνεχίζουν να διατίθενται με παράνομο τρόπο και συνεχίζουν να κυκλοφορούν και εκτός των Ιταλικών συνόρων. Εγώ προέρχομαι από μια περιοχή της Βόρειας Ιταλίας, το Βένετο. Ακόμα και σε αυτή την περιοχή, πολύ συχνά εμφανίζονται απόβλητα που προέρχονται από άλλες περιοχές, από αυτές δηλαδή που ανέφεραν οι αναφερόμενοι, οι συντάκτες της αναφοράς. Αυτό το σύστημα των αποτελεσματικών πρέπει να το αλλάξουμε. Η Κομισιόν πρέπει να το καταλάβει, αλλά ακόμα και το Προκοινοβούλιο. Πρέπει να υπάρξει παρέμβαση και με κανόνες και με νομοθεσία. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα ελέγχου που ξεπερνάει τον έλεγχο που ασκεί το εθνικό, τα εθνικά κράτη. Χρειαζόμαστε μια περιβαλλοντική αστυνομία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα που είναι η αιτία αυτού του προβλήματος είναι ότι στην Ιταλία, αλλά όχι μόνο στην Ιταλία, δεν υπάρχει στην πράξη η αρχή του ορυπαίνων πληρώνει. Στην Ιταλία είναι αδύνατον να βρει κανείς τον υπεύθυνο. Αν πάμε να δούμε τις καταδίκες που δόθηκαν στους υπέτειους αυτών, αυτής της μόλυνσης, δεν υπάρχουν πουθενά, δεν υπάρχουν καταδίκες. Το σύστημα δεν λειτουργεί. Δεν χρειάζεται λοιπόν ευρωπαϊκή νομοθεσία, ούτως ώστε να βοηθηθούν αυτά τα κράτη-μέλη που είτε διαφορούν ή δεν έχουν την δύναμη ή έχουν τρομακτικές αντιστάσεις μέσα τους που δεν μπορούν να τις ξεπεράσουν. Δεν, δεν πρέπει να έχουμε έναν κανόνα, μία νομοθεσία που θα εξασφαλίζει το ορυπενον πληρώνει. Ακόμα και στην δική μου την περιοχή, στην βορειοανατολική Ιταλία, τα ίδια προβλήματα έχουμε την καμπάνια. Έχουμε περίπτωση α, ρήπανσης, ε, περίπτωσης ρήπανσης απίστευτων διαστάσεων μολύνεται ο υδροφόρος ορίζοντας χωρίς, κανά, χωρίς καμία επίπτωση. Κανένα δεν ε, τιμωρείται. Πρέπει να υπάρχουν κυρώσει, να υπάρχει σιγουριά ότι θα υπάρξουν κυρώσει. Ό,τι αφορά την ανιχνευσιμότητα των αποβλήτων, και εδώ δυστυχώ πρέπει να πω ότι υπήρχε ένα σύστημα που είχε δρομολογήσει η Ιταλία, το λεγόμενο σύστρι, ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή που προέβλεπε την ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τον ηλεκτρονικό εντοπισμό των απορριμμάτων αλλά από αυτά που μάθαμε πριν από τρει-τέσσερι μήνε, προέκυψε ακόμα ένα από τα κλασικά ιταλικά σκάνδαλα. Δηλαδή, υπήρχε μια επιχείρηση που θα έφτιαχνε αυτό το ηλεκτρονικό σύστημα. Ε, έγινε διαγωνισμός με προσφορές ε, διογκωμένες, ε, παρενέβη αστυνομία, έγιναν συλλήψεις. Ακόμα και αυτό το, αυτή τη σημαντική απόπειρα την τρομολογήσαμε, αλλά τελικά ήταν θνησιγενή. Πέθανε το γεννάστε. Νομίζω ότι η Επιτροπή σα πρέπει να παρέμβει. Πρέπει να στραφεί προ την Κομισιόν για να υπάρξει τέλο πάντων μια κάποια δράση. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε στην ίδια τραπό που ακολουθήσαμε μέχρι στιγμή, γιατί δεν είχαμε καμία βελτίωση. Να αλλάξουμε στρατηγική. Ευχαριστώ. Grazie. Και εγώ ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Άλλος κανείς ζητά το λόγο. Mm, Όχι, δεν υπάρχει άλλο. Να πω και εγώ δύο λόγια τώρα. Ή μάλλον να απευθύνω κάποιε ερωτήσει προ την Κομισιόν, προ τον κύριο Μαγκανάρο. Η Κομισιόν λέει ότι έχει ξεκινήσει μια διαδικασία επί απέναντι στην Ιταλία. Από ό,τι ξέρω όμως, σε αυτή την αιτιολογημένη έκθεση που συνέταξε η Κομισιόν για αυτή τη διαδικασία, δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη αναφορά στο ειδικό αυτό πρόβλημα που αναφέραμε και που ακούσαμε. Το 2010 και 2011 ξεκίνησε μία διαδικασία επιπαραβάση κατά της Ιταλίας γιατί δεν σεβάστηκε την οδηγία για και σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά αδικήματα. Τι έγινε με αυτή τη διαδικασία που είχε ξεκινήσει το 2011. Έκλεισε. Η Ιταλία συμμορφώθηκε. Με τα όσα επιτάσσουν ε, τα ευρωπαϊκά κείμενα για τα περιβαλλοντικά αδικήματα. οι αναφερόμενοι ζητούν να, εφαρμοστεί η οδηγία 35 του 2004 σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική ευθύνη. Αυτή την έννοια τα ανέφεραν πολλές φορές οι Ιταλοί που πήραν το λόγο. Η Ιταλία και το Ιταλικό σύστημα δεν εφάρμοσε σωστά την σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Τι κάνει η Κομισιόν. μας παραπέμπει το θέμα στο δικαστήριο. Ένα ακόμα θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως συνέβη με την Ιταλία, με την Ελλάδα, με την Ισπανία, όταν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα, μπορεί να υποκαταστήσει α, τη δράση των κρατών μελών. Όταν δεν μπορούν να δράσουν οι εθνικές αρχές λόγω κρίσης, λόγω φτώχειας, ε, στέλνει δεκάλογους, στέλνει κανόνες που πρέπει να ακολουθήσουν τα εθνικά κράτη α, επειδή ακριβώς δεν κάνουν τίποτα. Όταν έχουμε τέτοιες παραβιάσεις της νομοθεσίας, που αφορούν την υγεία των πολιτών. Μπορεί η Κομισιόν να συνεχίζει να δράμα αυτόν τον τρόπο. Μιλάμε για παραβιάσεις εναντίον της υγείας των πολιτών, του περιβάλλοντος στο οποίο ζουν οι πολίτες. Μιλάμε για αξίες πολύ πιο σημαντικές από τις οικονομικές αξίες. Ίσως η Κομισιόν θα πρέπει να κατέβει πιο δυναμικά, αγνοώντας ε, έστω το, το θέσφατο της ε, αρχής της επικουρικότητας θα πρέπει να κάνει κάτι πιο δυναμικό, να παρέμβει πιο αποφασιστικά. Ε, δεν ξέρω αν θέλει να πει κάτι η Κομισιόν, τόσο ώστε να ενισχύσουμε έτσι, με την παρέμβαση της Κομισιόν την έκθεση. Εν θερμό δεν μπορώ να παρέμβω. Σε ό,τι αφορά τελευταία σας αυτή παρατήρηση, είναι αλήθεια ότι σε ορισμένου τομεί η Κομισιόν έχει πολύ πιο αποφασιστικές αρμοδιότητες. Θερυπή στο τομέα του ανταγωνισμού, ναι. Η Κομισιόν εκεί μπορεί απευθείας να επιβάλλει χρηματικές ποινές, χρηματικές κυρώσεις, όταν θεωρείται ότι παραβιάζει την νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, αλλά στο περιβα... σε ό,τι αφορά την νομοθεσία για το περιβάλλον, δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα. Δεν έχουμε τέτοιε αρμοδιότητε, τόσο έντονε αρμοδιότητε σε ό,τι αφορά το περιβάλλον. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει η Κομισιόν, αν οι αρμόδιε αρχέ δεν διαχειρίζονται επαρκώς σωστά την κατάσταση είναι να εκινήσει μια διαδικασία επί παραβάση. Αυτή τη στιγμή ξεκινήσει αυτή η διαδικασία και αν οι εθνικές αρχές συνεχίζουν να μην συμμορφώνονται, το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει η Κομισιόν είναι να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να ε, αποφανθεί και να καταδικάσει το κρατός μέλος. Εάν όντως υπάρξει καταδίκη, τότε δίδεται δίκιο στην ε, Κομισιόν αν ας πούμε κάνει μία σύσταση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, πάντα ε, παραπέμπουμε το θέμα στις ε, εθνικές αρχές και αυτές πρέπει να δράσουν. Δυστυχώς αυτό επιτάσσουν οι συνθήκες. Μπορούμε να τροποποιήσουμε αυτό το σύστημα, αλλά πρέπει για να το κάνουμε να τροποποιήσουμε τις συνθήκες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα συγκεκριμένα ερωτήματα που μου θέτετε, αν κατάλαβα καλά αυτά που μου είπατε, Θες να μάθετε αν η σημερινή ε, διαδικασία επί για το πρόβλημα της καμπάνιας αφορά και τα ειδικά βιομηχανικά απόβλητα. Αυτό ήταν το ερώτημά σας. Όχι. Απλώς έκανα μια παρατήρηση σχετική, ότι μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας επί δεν υπάρχει κάτι το ειδικό σε σχέση με, τα, με τις ειδικές καταγγελίες που ακούσαμε σήμερα. Δεν υπάρχει μια ειδική αναφορά. Μιλάμε για ειδικά απόβλητα, για επικίνδυνα απόβλητα που θα πρέπει να τα αντιμετωπίσει διαφορετικά η νομοθεσία από ό,τι τα συνήθη απόβλητα. Ναι, όντως δεν καλύπτουμε ε, στη διαδικασία αυτή τα ειδικά απόβλητα. Αλλά όντως, στα πλαίσια των επαφών που έχει η Κομισιόν με τις Εθνικές Αρχές, ζήτησε η Κομισιόν από τις ε, Ιταλικές Αρχές να εξασφαλίσουν μια σωστή διαχείριση και των ειδικών αποβλήτων. Θεωρεί ότι είναι δικό τους καθήκον. Όπως είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση, η Κομισιόν ζήτησε επίσης από τις Ιταλικές Αρχές να υιοθετήσουν ένα σχέδιο διαχείρισης για τα ειδικά απόβλητα στην καμπάνια, πέρα από το σχέδιο που έχουν υιοθετήσει για τα αστικά απόβλητα. Σε ό,τι αφορά τη σωστή εφαρμογή στην Ιταλία τη οδηγία για τα περιβαλλοντικά δικήματα, από ό,τι ξέρω δεν υπάρχει σχετική διαδικασία παραβάση που έχει ξεκινήσει. Η υπηρεσία μου δεν ασχολείται άμεσα με το θέμα αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν συνάδελφοι που επαληθεύουν τη σωστή εφαρμογή αυτής της ε, οδηγίας στην εσωτερική νομοθεσία όλων των κρατών μελών. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ανοιχτή διαδικασία επί παραβάση εναντίον της ε, Ιταλίας. Σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή της οδηγίας για την παραγωγική ευθύνη υπάρχει μια διαδικασία κατά της Ιταλίας. Η Κομισιόν δηλαδή θεωρεί ότι η Ιταλία δεν έχει εφαρμόσει σωστά όλα τα άρθρα της ε, σχετικής αυτής οδηγίας. Και αυτή η, παράβαση, η διαδικασία επιπαραβάση είναι στη φάση της ε, αιτιολογημένης ε, έκθεσης. Γνώμης. Και αν δεν συμμορφωθεί η Ιταλία θα πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Σας ευχαριστώ. Νομίζω λοιπόν ότι μπορούμε να κλείσουμε τη συζήτηση σε αυτές τις αναφορές. Το αίτημα όλων είναι να μείνουν ανοιχτές αυτές οι αναφορές. Ο κύριος Γιάρ έκανε το εξής αίτημα, να έρθουμε ξανά σε επαφή με τις αρμόδιες Ιταλικές αρχές και να επαναδιατυπώσουμε εξ ονόματος της Επιτροπής Αναφοράς την πρόσκληση, την πρόσκλησή μας προς την ε, Ιταλική κυβέρνηση και, το, και προς τα αρμόδια Υπουργεία, προς τα οποία έχουμε ήδη απευθυνθεί στο παρελθόν, να παρέμβουν εκ νέου, ούτω ώστε να κάνουν αυτό που οφείλουν να κάνουν. Ο πρόεδρος της ε, περιφέρειας έχει ειδική αρμοδιότητα σε σχέση με την έγκριση και την εφαρμογή του σχεδίου για τα αστικά απόβλητα και τα ειδικά απόβλητα που είναι δύο διαφορετικά σχέδια. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι θα, κάνω, θα προσθέσω και μία ακόμα έκκληση. Μία έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ανασκουμποθεί περισσότερο, να παραπέμψει την Ιταλία για περιβαλλοντικά δικήματα. Η διαδικασία που έχουμε ξεκινήσει αφορά την ε, περιβαλλοντική ευθύνη της Ιταλίας. Είναι μια άλλη διαδικασία. Ε, επ' αυτής μπορούμε σήμερα να δράσουμε. Για αυτή τη διαδικασία ζητάμε από την ε, Κομισιόν περισσότερες λεπτομέρειες, περισσότερα στοιχεία, μια μεγαλύτερη και πιο δυναμική παρέμβαση. Απλό, να μην ξεκινήσει έτσι απλώς μια διαδικασία επί παραβάση για τη διαχείριση, όπως αυτή που ξεκίνησε για τη διαχείριση των αποβλήτων στην καμπάνια, αλλά μια νέα διαδικασία για την άλλη πλευρά του δράματος που ζει αυτή τη στιγμή η καμπάνια. Τώρα, από πλευράς μας μπορούμε ίσως να υποβάλουμε ένα ερώτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή εμείς ως Επιτροπή Αναφορών υποβάλλουμε ένα ερώτημα σχετικό με το θέμα αυτό προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα το θέσω αυτό το θέμα και στους συντονιστές. Εάν συμφωνείτε, κλείνουμε εδώ τη συζήτηση για αυτές τις δύο αναφορές. Ευχαριστώ τους συντάχτες των αναφορών αυτών που ήρθαν εδώ. Θα τους ενημερώσουμε για τις εξελίξεις. Και τώρα θα περάσουμε στην αναφορά που εμφανίζεται στο σημείο 7 της ημερησίας διάταξης. Είναι η αναφορά του Φαμπιάνο Φιλιππίν, Ιταλικής Ιθαγένειας, φέρουσα τέσσερις υπογραφές, σχετικά με την παρουσία ασυνήθιστων ποσοστών διοξίνης σε ζώα ελευθέρας βοσκής στο Φριούλι, σε μια συγκεκριμένη περιοχή του Φριούλι. Θα μας παρουσιάσει αυτή την αναφορά ο κύριος Φαμπιάνο Φιλιππίν είναι εδώ στην αίθουσα. Θα του δώσω το λόγο για πέντε λεφτά. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μιλήσω στα Ιταλικά. Παρακαλώ, παρακαλώ, κυρία Όκεν, μπορείτε να βγείτε έξω. Ε, ευχαριστώ, θα μιλήσω Ιταλικά. Σας ευχαριστώ για την προσοχή. Σας ευχαριστώ που ήρθατε να ακούσετε ένα πρόβλημα που μας απασχολεί όλος ιδιαίτερος. Έφτασα πέντε λεφτά νωρίτερα. Αυτό ήταν χρήσιμο. Και για, το, και για μένα και για το φίλο μου, τον κύριο Ρατζανόνη, που ασχολούμαστε με τα προβλήματα, τα περιβαλλοντικά στην επαρχία μου. Ε, έτσι λοιπόν θα, θα μιλήσω για ένα θέμα που συνδέεται με αυτά που ακούσατε για την καμπάνια. Θα σας δώσω εγώ ένα άλλο παράδειγμα για να σας παρουσιάσω καταρχάς το πρόβλημα στο Φριούλι. Υπάρχει μια άλλη περιοχή, στον Τάρανδο, που ζει ανάλογο πρόβλημα με εμά. Μιλάμε για πρόβλημα που εμφανίζεται σε μια περιοχή βιομηχανική, που γειτονεύει όμως με αγρούς και χωράφια. Έχουμε χημικά εργοστάσια, χημικές βιομηχανίες, αλλά πολύ κοντά έχουμε χωράφια. Δημιουργούνται προφανώς προβλήματα στους μήκητες στις αναπνευστικές οδούς των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιοχή. Ο κύριος Τζανόνι που ακούσατε πριν μας ξέρει πολύ καλά με συμμετείχε σε μία σειρά από συνέδρια που οργανώσαμε για το πρόβλημα αυτό και άκουσε το πρόβλημα. Ε, δυστυχώς οι Ιταλικές αρχές συνεχίζουν τη γνωστή τους αδιαφορία. Είμαι νομικός. Συμμετείχα σε διάφορες επιτροπές ε, που συζήτησαν αυτό το πρόβλημα. Πριν από 50 χρόνια είχαμε αντίστοιχα τραγικά γεγονότα. Εγώ ως ε, Δημοτικός Σύμβουλος ε, ζήτησα να γίνει μία μελέτη για να καταλάβουμε ποια είναι τα εδάφη στην Ιταλία που είναι ασφαλή και ποια είναι τα δηλητηριασμένα. Μέχρι στιγμής δεν έγινε αυτή η μελέτη. Έγινε μια επιδημιολογική μελέτη για να δούμε εδώ και 5 ή 6 δεκαετίες ε, ποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην υγεία τους και στο DNA τους λόγω της μόλυνσης στην περιοχή μας. Τίποτα δεν έγινε. Ε, μετά από ε, διάφορα συνέδρια, κάναμε κάποιες αναλύσεις σε κοτόπουλα. Ο κύριος Τζανάνη συμμετείχε για αυτό το συνέδριο για το Μανιάγκο, την περιοχή αυτή που σας παρουσιάζω. και κάναμε αυτή την, ε, ένα πείραμα σε ε, κοτόπουλα, τα οποία μας είπαν ότι μάλλον είχαν, φάει ε, μολυσμένη τροφή από μπάρμπεκιου. Ο κ. Κανέλη από το Τριβένετο ε, συμμετείχε σε μία, σε μία έκθεση, σε μία μελέτη που έγινε ο κύριος Κανέλη ε, σε αυτή την έκθεση είχε παρουσιάσει και κάποιες φωτογραφίες πολύ αποκαλυπτικές ε, που δείχνουν ότι σε όλα τα τρόφιμα ε, που ελέγξαμε το 2010 και 2011, σε όλα τα τρόφιμα, μιλάμε για κοτόπουλα, μιλάμε για κρέας από, ε, και κόκκινο κρέας ας πούμε, υπάρχει διοξίνη κάναμε αυτή την ανάλυση. Ξέρετε ότι αυτές οι αναλύσεις είναι πολύ ε, δαπανηρές. 200 ευρώ κοστίζει η ανάλυση στο κοτόπουλο και όμως σήμερα ε, λόγω κρίσης ε, δεν υπάρχουν χρήματα για να γίνουν τέτοιου είδους αναλύσεις που είναι δαπανηρές. Αλλά αυτό δεν μπορεί να είναι δικαιολογία. Η κατάσταση που σας παρουσιάζουν είναι πάρα πολύ σοβαρή. Σας ευχαριστώ που με ακούτε. Εσείς θέλω να με ακούσετε, διότι από τις Ιταλικές Αρχές μέχρι στιγμής είχαμε μικρή ανταπόκριση. Καταλήγοντας, θα ήθελα να κάνω μία πρόσκληση. Θα ήθελα να έρθετε στην περιοχή μας. Άκουσα πριν την κυρία Όκεν, η οποία μίλησε για μια επίσκεψη που κάνατε στην Ιταλία για τα απόβλητα στην Νάπολη. Εάν έρθετε στο Μανιάγκο, σε αυτή τη μικρή πόλη, που δυστυχώς δεν εμφανίζεται σε, στις ειδήσει γιατί έχει πολύ λίγο κόσμο, πολύ λιγότερο από τον Τάραντο. Τον Τάραντα, συγγνώμη. Ε, θα καταλάβετε ποιο είναι το πρόβλημά μας. Δυστυχώς υπάρχει μεγάλη διαφορία για το πρόβλημά μας. Ε, καλό θα ήταν για να, να έρθετε για να κάνετε ένα μικρό πείραμα. Ο κ. Τζανόνι έχει δίκιο ότι στην Ιταλία ε, είναι δύσκολο να βρεις τους υπεύθυνου. Εγώ είμαι δικηγόρος και το ξέρω. Ε, συμμετείχα σε πολλές περιβαλλοντικές επιτροπές και συχνά για αυτά τα δικήματα υπάρχει παραγραφή. Πέρασε υποτίθεται πολύ καιρό και είναι πολύ δύσκολο να βρούμε του υπεύθυνου για το κάθε έγκλημα. Δεν θα θέλαμε στο Μανιάγο να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί η κατάσταση αυτή ε, εξελίσσεται εδώ και πολλά χρόνια και τα οι αρνητικέ επιπτώσεις πάνω στον περιβάλλον και στον πληθυσμό είναι εμφανεί κάθε μέρα. Κλείνω. Ε, ελπίζω να μην ξεπέρασα τα πέντε λεπτά. Υπάρχουν εκτός από αυτή την αναφορά και άλλες αναφορές παρόμοιες, ε, με παρόμοια προβλήματα με αυτά που σας ανέφερα. Αυτά και σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για την παρέμβασή σας. Τώρα θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της ε, Κομισιόν. Thank you uh, for giving me the floor. So... Ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Σε ό,τι αφορά την βιομηχανική περιοχή Μαγκιάνα και γενικότερα την περιοχή του Φριούλη φύσταται κοινωτική νομοθεσία που ε, εφαρμόζεται και η Κομισιόν δεν έχει διαπιστώσει παραβίασή της προς το παρόν. Συνεπώς δεν έχει αναλυθεί κανόνας είδους δράση από πλευράς Κομισιόν. Αυτό επιβεβαιώθηκε και από τις Ιταλικές Αρχές που αναφέρουν, ανέφεραν ότι το Περιφερειακό Γραφείο Προστασίας του Περιβάλλοντος, το ΆΡΠΑ, διενήργησε αναλύσεις εκπομπών αλλά και ειζημάτων διοξίδι, ε, διοξίνης ε, και PCB ε, κοντά, ε, ανάντι και κατάντι της ε, τσιμεντοβιομηχανίας και οι τιμές οι οποίες ανοιχνεύθησαν δεν υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια που προβλέπει η νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά τα υψηλά επίπεδα διοξίνης στα κοτόπουλα ελεύθερης βοσκής, θα ήταν χρήσιμο να δούμε τις λεπτομέρειες της ανάλυσης στην οποία αναφέρεστε, διότι δεν γνωρίζουμε ποια είναι η τιμή η οποία ανοιχνεύτηκε πάντως ε, σίγουρα προφανώς θα πρέπει να υπερεύαιναν οι τιμές αυτές που καθορίζει ο κανονισμός 81 του 2006. Ε, σε αυτή την περίπτωση θα έπρεπε να ξεκινήσει μια έρευνα προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα αίτια. Ε, οι Ιταλικές αρχές από την άλλη μεριά μας ενημέρωσαν ότι πέραν αυτού του κρούσματος, των κοτόπουλων δηλαδή, δεν έχουν ανοιχνεύσει κανένα είδου άλλη παράβαση, υπέρβαση ορίων της κοινωτικής νομοθεσίας. Παρ' όλα αυτά, μας ενέφεραν ότι παίρνουν πολύ στα σοβαρά το θέμα και προσπαθούν να εντοπίσουν την πηγή του προβλήματος προκειμένου να ε, διαπιστώσουν αν το πρόβλημα συνδέεται με την βιομηχανία, με το εργοστάσιο. Ε, Ιδιαίτερως προσπάθησαν να εντοπίσουν ζώα στην περιοχή που τρέφονται με ντόπιε ζωοτροφές ε, αποκλειστικά ντόπιε ζωοτροφές. Όμως δεν βρήκαν τέτοια αγροκτήματα δεν βρήκαν τέτοιες εκμεταλλεύσεις που να ε, δίνουν στα ζώα τους μόνο ντόπιε ζωοτροφές. Οπότε δεν προκύπτει άμεση σύνδεση με, την, ε, το εργοστάσιο. Πλην όμως οι τελικές αρχές ε, διενεργούν αυτή τη στιγμή, έχουν θέση μάλλον σε εφαρμογή ένα πιο πλήρες σχέδιο δειγματοληψίας προκειμένου να εντοπιστούν να εντοπιστεί η πηγή. Ε, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα αυτό το project, θα ξεκινήσει επόμενε εβδομάδε. αλλά αυτή τη στιγμή οι Ιταλικές αρχές δεν γνωρίζουν καμιά ε, περίπτωση παράβασης, πλην όμως θα ερευνήσουν τα υψηλά επίπεδα διοξίνης και θα διαπιστώσουν το κατά πόσον αυτά συνδέονται με την ύπαρξη εργοστασίου στην περιοχή. Η Κομισιόν θα παρακολουθήσει τη δράση των Ιταλικών αρχών ε, και έχουμε ζητήσει τακτική ενημέρωση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το πρόβλημα αυτό δεν αφορά μόνο τη συγκεκριμένη περιοχή. οι αναλύσεις που έγιναν δίνουν περιεκτικότητα σε διοξίνη πολύ ψηλότερη από την ε, ε μέγιστη επιτρεπόμενη. η αιματοληψία έγινε σε διάφορες περιοχές οι οποίες είναι μολυσμένες. Θα πρέπει να θέσουμε το εξής ερώτημα. Μήπως θα έπρεπε να ε, διαχωρίσουμε γεωγραφικά τις ε, περιοχές, τις βιομηχανικές περιοχές από τις περιοχές ε, στις οποίες επιτρέπεται να εκτρέφονται ζώα για ανθρώπινη κατανάλωση. Στην Πρέσια, στην Ιταλία, έχουμε για παράδειγμα ένα αποτεφρωτήριο το οποίο λειτουργεί εδώ και αρκετά χρόνια και που ποτέ δεν ξεπέρασε τα μέγιστα επιτρεπόμενα όρια εκπομπών όπως προβλέπονται από τους κανονισμούς. Όμως, όμως στην γειτονική περιοχή κλείσαμε προληπτικά όλες τις εκμεταλλεύσεις ε, τροφές ε, αγελάδων και βοηδών της περιοχής γιατί είχε ανοιχνευτεί ψηλό επίπεδο διοξίνης. Συνεπώς ε, υπάρχουν κανόνες ε, που απαγορεύουν την υπέρβαση συγκεκριμένων μέγιστων εκπομπών, αλλά αυτό δεν αποτελεί πάντοτε εγγύηση. Πολλές φορές βλέπουμε συσσόρευση μολυσματικών ουσιών ε, στο χώμα. Τα ζώα μπορούν βοσκώντας να ε, πάρουν ένα τμήμα αυτών των ουσιών το οποίο τελικά μπορεί να καταλήξει στο γάλα και μάλιστα και στο γάλα το οποίο ε, φτάνει στις μητέρες και γίνεται μητρικό γάλα. Οι αναλύσεις που έγιναν κοντά στον αποτεφρωτή έδειξαν ότι οι θυλάζουσες μητέρες ε, ε, δίνουν και αυτές υψηλά επίπεδα διοξίνη στο γάλα τους. Με λίγα λόγια παράγουν γάλα μολυσμένο ε, με διοξίνη. Το χημείο μας, το χημείο του κράτους, επιβεβαίωσε ότι η νομοθεσία δεν είναι επαρκής ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο κοκτέιλ, έτσι το ονομάζουν. Ο Επίτροπος Ποτόσνικ, μάλιστα, ανέφερε ότι στην κοινωνική νομοθεσία δεν προβλέπονται ελάχιστες αποστάσεις ε, ιατρικών μονάδων εκμεταλλεύσεων από ε, τέτοιου τύπου ε, εγκαταστάσεις όπως οι αποτεφρωτές. ή, οι εγκαταστάσεις κάψεως. Εμείς στην Ιταλία έχουμε ένα διεθνώς αναγνωρισμένο και πιστοποιημένο εργαστήριο, χημικό εργαστήριο, που εντόπισε μάλιστα και τις ε, διοξίνες στην Μπρέσια και στα κοτόπουλα του Μανιάγο και τις διοξίνες στο γάλα το, στο μητρικό γάλα. Αυτό το εργαστήριο λοιπόν έκανε όλες αυτές τις ε, ανακαλύψεις, αλλά χρειάστηκε να κλείσει διότι η περιοχή του Βένετο του μείωσε τον περιπολογισμό, μείωσε και δεν μπορεί να το χρηματοδοτήσει πια. Η Ευρωπαϊκή ε, το Ευρωπαϊκό Γραφείο Ασφάλειας των Τροφίμων θα έπρεπε να ερευνήσει λοιπόν και αυτές τις περιπτώσεις, να κάνει μια ε, επιστημονική έρευνα και να προτείνει ενδεχομένω ε, νομοθεσία για προστατευόμενες περιοχές όπου, ε, που επειδή είναι κοντά σε βιομηχανικές μολύνσεις, βιομηχανικές μονάδες να μην επιτρέπεται να μην επιτρέπονται κτηνοτροφικές δραστηριότητες ε, ή γεωρικές δραστηριότητες. Ενδεχομένως επίσης θα έπρεπε να τροποποιηθούν και τα μέγιστα όρια μολυσματικών παραγόντων στο έδαφος. Όπως είπε και ο αναφερόμενος, οι τοπικές αρχές δεν βοηθάνε ε, στη διαφώτιση του φαινομένου. Στην πράξη, ό,τι αποκαλύπτεται οφείλεται σε εθελοντικές ε, πρωτοβουλίες της τοπικής κοινωνίας και τοπικών οργανώσεων. Έτσι μόνο ε, εντοπίζονται αυτά τα προϊόντα τα οποία έχουν μολυνθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Μποστινάρου. Ευχαριστώ. Δυο λόγια μόνο. Νομίζω ότι είναι σημαντικό και εδώ να λάβουμε υπόψη το σορευτικό αποτέλεσμα. Γιατί η συνεχιζόμενη επίμονη μόλυνση μέσα από διάφορους τρόπους κυρίως με υψηλή τοξικότητα στοιχεία και λαμβάνοντας υπόψη το σωρευτικό τους αποτέλεσμα, δημιουργούν δραματικές επιπτώσεις στην κατάσταση της υγείας του πληθυσμού που ζει στις παρακείμενες περιοχές. Και είναι σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εδώ να ζητήσει από τις αρμόδιες αρχές κάποια στιγμή να αξιολογήσουν το σωρευτικό αποτέλεσμα της επίμονης μόλυνσης στην υγεία του πληθυσμού. Γιατί μόνο αν δούμε τις επιπτώσεις στο νερό, έδαφος, αέρα, θα πάρουμε ένα κομμάτι της αλήθειας, αλλά όχι ολόκληρη την αλήθεια. Και δεν θα έχουμε ένα μακροπρόθεσμο ε, στοιχείο Δηλαδή δεν θα δούμε τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που αυτές είναι καθοριστικές για την υγεία του πληθυσμού. Εδώ υπάρχει ένα ξεκάθαρο κενό στην ενωσιακή νομοθεσία. Η Γενική Διεύθυνση για το Περιβάλλον μιλάει για σωρευτική επίπτωση ή αντίκτυπο, αλλά αυτή είναι μια ε, λέξη μόνο, χωρίς περιεχόμενο, προκειμένου περί πρακτικής εφαρμογής και μετρήσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Κανείς άλλος δεν ζητεί το λόγο νομίζω. Οπότε αφήνουμε ανοιχτή την αναφορά και θα περιμένουμε τι θα απαντήσουν και οι εθνικές αρχές γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ενημέρωσε ότι περιμένει πληροφορίες αφού τη ζήτησε από τις Ιταλικές αρχές. Περιμένουμε λοιπόν. και θα κάνουμε και εμείς ίσως έτοιμα από την Επιτροπή μας απευθυνόμενοι στις περιφερειακές και τοπικές αρχές ε, για να στηρίξουμε αυτή την υπόθεση. Δεν νομίζω να κάνουμε τίποτα άλλο, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ίσως να συνεργαστούμε και με την Επιτροπή Περιβάλλοντος και να στηρίξουμε το έργο της Επιτροπής Περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τις νομοθετικές δραστηριότητες και την κατάρτιση της οδηγίας. Δεν νομίζω να μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Λοιπόν, κλείνουμε τη συζήτηση τώρα για αυτή την αναφορά, υιοθετώντα αυτή τη θέση. Εντάξει, εντάξει. Σας ευχαριστώ. Αυτό Λοιπόν, έχουμε και μία ακόμη αναφορά. Στο σημείο 8. Είναι η αναφορά του κυρίου Ζαν Πυρότ. Ο κύριος Ζαν Πυρότ είναι εδώ. Έχετε το λόγο για πέντε λεπτά. Η αναφορά μου αφορά τον χρόνο εργασίας των εθελοντών πυροσβεστών. Γνωρίζουμε ότι η κοινωτική νομοθεσία υπερισχύει της εθνικής νομοθεσίας και παραβιάζεται όταν ένα κράτος όπως το Βέλγιο ή Γαλλία θεωρεί ότι ένας εργαζόμενος που έχει προσληφθεί ε, ως πυροσβέστης ε, είναι απλώς ένας εθελοντής ενώ στην πραγματικότητα ε, έχει υπηρεσιακή κατάσταση και εργάζεται στο πλαίσιο ε, σύμβασης εργασίας περιορισμένης διάρκειας και κάνει την ίδια δουλειά που κάνουν και οι υπόλοιποι επαγγελματίες συνάδελφοι του. Γνωρίζουμε ότι το κοινοτικό δίκαιο ορίζει τον εργαζόμενο στο άρθρο 3 της Οδηγίας 89-391 ως οποιοδήποτε άτομο ε, εργαζεται για έναν εργοδότη όπως και οι μαθητευόμενοι και οι φοιτητές στα μαθητείας εκτός του οικιακού προσωπικού. Άρα λοιπόν περιλαμβάνονται οι ε, πυροσβέστες. Αυτή η οδηγία ε, συμπεριλήφθηκε στην 2003 του 88 μέσω του ε, άρθρου 1, σημεία 3 και 4 και της αιτιολικής έκθεσης. Γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι στον ειδικό και τον δημόσιο τομέα και οι πυροσβέστες ε, εργάζονται 168 ώρες μηνιαίως στην υπηρεσία τους αυτοί οι υπάλληλοι ε, κατά τη διάρκεια του έτους ε, εργάζονται ε, κατά μέσο όρο 70 ώρες την εβδομάδα για περίοδο 4 μηνών αντί για 48 ώρες όπως η αναφέρει η Οδηγία 2003 το 88 η οποία δεν προβλέπει και εξαιρέσεις. Η λέει ότι η βελτίωση της ασφάλειας υγιεινής και της υγείας των εργαζομένων στο χώρο εργασίας αντιπροσωπεύει έναν στόχο ε, ο οποίος ε, δεν μπορεί να ε, πληγεί από οποιαδήποτε, οποιαδήποτε οικονομικό σκεπτικό. Η εγκύκλειος του Βελγικού Υπουργείου Εσωτερικών του 2008 επιτρέπει στους εργοδότες δύο δυνατότητες. Ή ε, επιβάλλει ε, στους ε, πυροσβέστες τη, τον, τη βάρδια σε συγκεκριμένο πυροσβεστικό σταθμό ή, στην, ή τους επιβάλλει βάρδια στην περιοχή στην οποία εργάζονται. Και στις δύο περιπτώσεις τους, είναι προφανές ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται εκεί που του ζητάει να βρίσκεται ο εργοδότης. Και είναι έτοιμοι να αντιδράσουν σε όταν του ζητηθεί. Είναι προφανώς, προφανώς λοιπόν ότι η παραμονή τους εκεί εμπίπτει στο χρόνο εργασίας ε, του, της ε, ε, απόφασης Τζέγκερ του 9 Σεπτεμβρίου 2003 οπότε του αφαιρείται το δικαίωμα που προβλέπει το άρθρο 2 του πρωτοκόλου 4 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ε, αν δεν ήταν αυτός ο χρόνος εργασίας, ε, τότε θα έπρεπε να θεωρείται ο χρόνος ξεκούρασης. Ε, οπότε δεν θα έπρεπε να έχει καμία υποχρέωση, τουλάχιστον καμία από τις υποχρεώσεις που θα του επιβάλλει ο εργοδότης του. Και στην λογική της οδηγίας 2003 του 88 δεν υπάρχει ενδιάμεση κατηγορία. Όλες οι θεωρίες μπορούν να θεωρηθούν ε, είτε χρόνος εργασίας είτε χρόνος ε, ξεκούρασης. Ε, δεν υπάρχει ενδιάμεση ε, κατηγορία. Ζητούμε λοιπόν εδώ και τρία χρόνια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, προσφύγει εναντίον του Βελγίου και οποιονδήποτε άλλων χωρών παραβιάζουν κατά τον ίδιο τρόπο την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία η οποία έχει ψηφιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να διορθώσει την κατάσταση ε, της, ε, ε κοινοποίησης των μελών της 6ης 5ης 2011. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ. Η κυρία Μάντλιν Ριντ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όπως εξήγησε ο αναφέροντας, πρόκειται για μια αναφορά όπου έχει ξεκινήσει η διαδικασία εδώ και καιρό ε, σε μια προφορική παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Επίτροπή το Δεκέμβριο του 2010, μίλησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επικοινωνήσαμε το Κοινοβούλιο το Μάιο του 2011. Ε, ο αναφέροντας έχει υποβάλει πρόσφατα παρατήματα στο Κοινοβούλιο το Μάιο και το Ιούνιο του 2013 και ετοιμάσαμε μια επιπλέον ανακοίνωση ε, προς απάντηση. Καταλαβαίνω ότι είμαστε στην ε, τελική φάση πριν διαβιβάσουμε το κείμενο αυτό στο Κοινοβούλιο. Βεβαίω δεν έχετε αυτό το κείμενο σήμερα στην Επιτροπή Αναφορών, αλλά πολύ σύντομα θα το λάβετε. Όπω σημειώνει και ο συντάκτη, στην τεκμηρίωσή του ε, έχει παράπονα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτό το θέμα, που ήταν αντικείμενο εκτεταμένη αλληλογραφία μεταξύ τη Κομισιόν και εκείνων. Η Κομισιόν έγραψε πολλέ φορέ στι εθνικέ αρχέ και υπήρξαν πάρα πολλέ δυσκολίε σε αυτήν την περίπτωση. Ήταν δύσκολο δηλαδή να βρούνε τα στοιχεία, τα αντικειμενικά, γιατί υπήρξαν πολλές αποφάσεις ε, τα προηγούμενα χρόνια από τα εθνικά δικαστήρια που άλλαξαν την ε, κατάσταση σε εθνικό επίπεδο. Τώρα, συγκεκριμένα για τα θέματα που θέτει η αναφορά, η αρχική αναφορά έθεσε θέματα που αφορούσαν τις αποδοχές. προκύπτει από τα στοιχεία ότι ο αναφέρον σε αυτό το στάδιο ασχολείται κυρίως με τα όρια του εργάσιμου χρόνου από την οδηγία ε, για λόγους υγείας και ασφάλειας. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τρία πράγματα που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση εδώ. Πρώτον, η αναφορά έχει να κάνει με τη λεγόμενη εθελοντική ε, εργασία στο Βέλγιο που καλύπτεται από την Οδηγία για τον Χρόνο Εργασίας και υπάρχουν και από το Δικαστήριο αποφάσεις σχετικά. Η θέση για τους εθελοντές πυροσβέστες και αν καλύπτονται από τις διατάξεις της οδηγίας είναι πιο σύνθετο θέμα. Το νομικό καθεστώς των εθελοντών πυροσβεστών διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, όπως και οι όροι υπηρεσία τους. Η θέση της Κομισιόν σε σχέση με αυτή την αναφορά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 20, ε, του 2011, είναι να ακολουθήσουμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που θεωρεί ότι ο ορισμός του, της εργασίας στην οδηγία για τον εργάσιμο χρόνο είναι ε, ορισμός ευρύς ε, και καλύπτει την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων με βάση το ενωσιακό δίκαιο και υπάρχουν κριτήρια που θα πρέπει να εφαρμόζονται από τα εθνικά δικαστήρια προκειμένου να κρίνουν εάν ο εργαζόμενος καλύπτεται από την οδηγία. Ο αναφέρον αναφέρεται στον ορισμό της οδηγίας για την υγεία και την ασφάλεια και το δικαστήριο αμφέβαλε αν ορισμός ισχύει για το, στην οδηγία για τον χρόνο εργασίας που εκεί είναι ο ορισμός που θα έπρεπε να εφαρμοστεί. Αυτό δεν είναι σημαντικό για την αναφορά αυτή, γιατί οι τελευταίες αποφάσεις του Βελγικού Δικαστηρίου ε, αναφέρουν ότι οι εθελοντές πυροσβέστες στα πλαίσια της υπηρεσίας στο Βέλγιο θα πρέπει να θεωρούνται ως εργαζόμενοι στα πλαίσια της οδηγίας και η Κομισιόν κινείται πάνω σε αυτή τη βάση. Το ερώτημα που προκύπτει από νομικής άποψης είναι η φύση του χρόνου που λαμβάνεται υπόψη για το σκοπό και για το, της αναφοράς. Ο αναφέρον ισχυρίζεται ότι ο χρόνος εργασίας και η περίοδοι ανάπαυσης των εθελοντών ε, πυροσβεστών δεν σέβονται τα όρια της οδηγίας γιατί εργάζονται ε, στη βασική δουλειά και προσφέρουν ως εθελοντές, πυροσβέστες και πρόσθετο χρόνο συμπληρωματικά. Πέρασε λίγος χρόνος για να καταλάβουμε πώς είχε ακριβώς αυτό το θέμα που είναι αρκετά περίπλοκο και να καταλάβουμε και καταλάβαμε μετά από εντελεχείς έρευνες ότι η θέση του βελγικού εθνικού δικαίου έχει ως εξή. Ο κανονικός χρόνος εργασίας που καλύπτεται από τους εθελοντές πυροσβέστες ήδη υπολογίζεται ως χρόνος εργάσιμος. όταν είσαι επιφυλακή και πρέπει να είναι παρόντος στον χώρο εργασίας που είναι κάποιο στρατόπεδο ή κάποιος χώρος και αυτός ο χρόνος ε, ε, ε, μετράει ως χρόνος εργασίας. Όταν όμως τους καλέσουν, όταν είναι στο σπίτι τους για να ανταποκριθούν σε κάποια κατεπίγουσα ανάγκη, ο χρόνος υπηρεσίας μέχρι να έρθουν από το σπίτι επίσης καλύπτεται και θεωρείται χρόνος εργασίας. Δηλαδή σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο ποσοστό, ο χρόνος αυτός ε, θεωρείται εργάσιμος χρόνος από τις εθνικές αρχές. Το ιδιαίτερο θέμα του αναφέροντος αναφέρεται σε μια ειδική μορφή υπηρεσίας, όπου οι αναφέροντες δεν είναι υποχρεωμένοι να παραμείνουν σε κάποιο χώρο, δηλαδή στις εγκαταστάσεις της πυροσβεστικής. Δεν, ε, να ε, ε, διανυκτερεύσουν εκεί, αλλά ε, καλούνται να παραμείνουν σε κάποια ακτίνα γύρω από τους εγκαταστάσεις. Μπορεί να μείνουν σε, στο σπίτι τους ή σε φίλους και είναι υποχρεωμένοι να μπορούν να, είναι, να, μπορούν να ανεβρίσκονται εύκολα, να μπορεί κανείς να επικοινωνήσει μαζί τους. Και ο χρόνος ο συγκεκριμένος για να ανταποκριθούν σε μια κλίση δεν είναι απόλυτα σαφής μετά από πότε πρέπει να αντιδράσουν. Από ό,τι αντιλαμβανόμεθα από τα διαθέσιμα στοιχεία είναι ότι μπορεί να είναι μέχρι 25 λεπτά και σε ορισμένε κοινότητε δεν υπάρχει καν χρονικό όριο. Ο αναφέρον λέει και μάλιστα στο τελευταίο παράρτημά του στην αναφορά του αναφέρει και μια εγκύκλιο υπουργική των εθνικών αρχών που φαίνεται να αναφέρει ότι ο χρόνος είναι μεταξύ τριών και πέντε λεπτών, δηλαδή πολύ λιγότερος. Ξέρουμε ότι κάποιε αποφάσει των εθνικών δικαστηρίων πάνω σε αυτό το θέμα αναφέρουν ότι ο χρόνο αντίδραση θα πρέπει να είναι 10 λεπτά, 1 τέταρτο. Και φαίνεται ότι διαφέρει ο χρόνο από κοινότητα σε κοινότητα. Σε σχέση με αυτό το τελευταίο λοιπόν που θέτει με την Υπουργική Εγκύκλιο Αναφέρον, ε, απευθυνθήκαμε και πάλι στι εθνικέ αρχέ, ζητώντα διευκρινήσει για το θέμα αυτό για να είναι απόλυτα σαφέ ότι θα μα δώσουν την ακριβή εικόνα τη κατάσταση, όπω ε, υπάρχει. Τώρα, σε σχέση με το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζεται από νομικής άποψης ο χρόνος αυτός. Η προσέγγιση της Κομισιόν στηρίζεται σε αυτό που αναφέρει ε, το δικαστήριο στις ε, αποφάσεις ΣΥΜΑΠ και ΓΕΓΕΡ. Η υπόθεση ΣΥΜΑΠ που αναφέρεται στους γιατρούς στην Ισπανία και στις εφημερίες τους κάνει κάποιες συγκεκριμένες διαφοροποίησεις μεταξύ του χρόνου που πρέπει να είναι ε, σε εφημερία στο χώρο εργασίας του οι γιατροί και στο χρόνο κατά τον οποίο πρέπει να είναι στη διάθεση της υπηρεσίας, αλλά μπορεί να είναι στο σπίτι τους και να έρθουν αν χρειαστούν. Η εφημερία θα πρέπει να θεωρείται, λέει το δικαστήριο, ως εργάσιμος χρόνος, αλλά η οδηγία λέει ότι όταν είναι ε, σε διαθεσιμότητα, ε, τότε αυτό δεν θεωρείται εργάσιμος χρόνος από την οδηγία. Το δικαστήριο αναφέρει και στην υπόθεση Γέγκερ την ανάλυση αυτή, Επίσης και αυτή είναι και η βάση για την νομική αξιολόγηση της Κομισιόν σχετικά με τον χρόνο εργασίας που αναφέρει ο αναφέρον. Τώρα, ε, θα πρέπει να έχουμε την απάντηση από τις βελικές αρχές για να διευκρινιστεί οριστικά το θέμα σχετικά με την ακριβή περίοδο κατά την οποία οι αθελοντές πυροσβέστες θα πρέπει να έχουν αυτό το χρόνο που θα είναι σε διαθεσιμότητα. Όμως η πρώτη μας αντίληψη είναι ότι αυτός ο χρόνος φαίνεται να είναι πολύ πιο κοντά στη διαθεσιμότητα που αναφέρουν τα δικαστήρια στις υποθέσεις ΕΜΑΠ και ΓΕΓΕΡ, όπου το δικαστήριο είπε σαφές ότι δεν θα πρέπει αυτός ο χρόνος να θεωρείται εργάσιμος βάσει της οδηγίας. Η πρόσθετη κοινοποίησή μας θα ασχοληθεί διεξοδικότερα με τα θέματα που αναφέρει ο αναφέρον και θα χαρώ να επανέλθω σε κάποια θέματα που μπορεί να θέσει η Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Α, συγγνώμη, λέει ο κ. Βουστινάρου, δεν, ε, δεν είμαι ευτυχής με την απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρώτον, είναι ασαφής ο ορισμός του τι είναι εργάσιμος χρόνος. Για ένα πυροσβέστη δεν υπάρχει δυνατότητα να ορίσουμε επακριβώς την διάρκεια του χρόνου εργασίας του. Θυμάστε την ε, ιστορία με τις φωτιές, τις πυρκαγιές στο Νιούαρκ, στη ΣΥΠΑ. Υπήρχε περιορισμός στο χρόνο εργασίας των πυροσβεστών τότε υπήρχε καμιά Αμερικανική αρχή που, τους έλεγε σταμάτα τώρα γιατί έληξε ο χρόνος εργασίας σου και από εδώ και πέρα θα πρέπει να αντικατασταθείς από άλλες ομάδες. Έγινε κάτι τέτοιο? Όχι, αφού δεν γίνεται. Δεν είναι, δεν είναι δυνατόν σε μεγάλες πυρκαγιές δεν υπάρχει η δυνατότητα να προβλέψει κανείς πόσο θα διαρκέσει η πυρκαγιά. Αυτό είναι μια ξεκάθαρη ιδιαιτερότητα ε, της πυροσβεστικής υπηρεσίας και του χρόνου εργασίας τους. Δεύτερον, τι γίνεται με τους εθελοντές και όταν παρεμβαίνουν αυτοί. Ον είναι, ας πούμε, μια μεγάλη πυρκαγιά Και μάλιστα τότε δεν είναι μόνο πυροσβέστες, μπορεί να παρέμβουν για να αντιμετωπίσουν καταστροφές, τρομοκρατική επίθεση. Ποιος θα πει ότι μετά από μισή ώρα και μετά από μία ώρα θα σταματήσει ο τρομοκράτης τη δουλειά του και θα σταματήσει και ο πυροσβέστης τη δικιά του τη δουλειά. Ποιος μπορεί να τα πει αυτά. Ε, δεν λέγονται αυτά, ε, οπότε υπάρχει θέμα ορισμού. Δεν λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητα της δουλειάς του πυροσβέστη. Δεύτερον, αυτοί είναι υποχρεωμένοι είτε να κάθονται σε κάποιον ιδιαίτερο χώρο, ειδικό χώρο, ή θα πρέπει να είναι στο σπίτι τους, αλλά έτοιμοι να αντιδράσουν σε πέντε λεπτά και τώρα δεν ξέρω ακριβώς μετά από ποιο χρόνο υποχρεούνται να πάνε στον χώρο που θα συγκεντρωθούν. Είναι σαν στρατός. Δεν μπορεί κανείς δηλαδή να αποφασίζει ελεύθερα και να λέει σήμερα ε, δεν έχω κανένα πρόβλημα να απαντήσω, αλλά αύριο γιορτάζω ή είναι μέρα γιορτής και δεν θα απαντήσω στην κλίση που δέχτηκα και θα βγάλουν πέρα μόνοι τους, χωρίς εμένα. Αυτή θα ήταν μια πολύ στενή ερμηνεία. Και οι πυροσβέστες δεν θα μπορούσαν να ε, δράσουν με την απαραίτητη αποτελεσματικότητα, είτε είναι εθελοντές είτε όχι. Από ό,τι φαίνεται, οι βελγικές αρχές, εν προκειμένου, δεν μπόρεσαν να περιγράψουν ακριβέστατα όπως πρέπει τις υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και των δύο πλευρών, και του εργοδότη και των εργαζομένων. Και να αποφασίσουν ποιος είναι ο χρόνος εργασίας και τι συμβαίνει αν οι άνθρωποι αυτοί συνεχίσουν να εργάζονται μετά την λήξη του χρόνου εργασίας που προβλέπει το βελγικό δίκαιο. Αν δηλαδή σταματήσει η δουλειά τους νωρίτερα μπορεί και να υποστούν κυρώσεις ε, ή να πάνε και στη φυλακή για, αν σταματήσουν πριν όμως ε, τελειώσει ε, πριν, πριν ε, πάυσει να υφίσταται η ανάγκη και πριν σβήσει η πυρκαγιά θα πρέπει οι βελγικές αρχές να μας δώσουν και άλλα στοιχεία, όλα αυτά που πρέπει να τα δει και να δώσουν και μια αξιοπρεπή απάντηση έτσι στον αναφέροντα. Εγώ δεν ξέρω τι απάντηση θα είναι αυτή αφού δεν είμαι και νομικός. Αλλά είναι προφανές ότι ο, ο, πυροσβέστης όταν κληθεί να πάει να κατασβέσει μια φωτιά θα πρέπει να είναι εκεί μέρα νύχτα, βρέξει χιονίσει. Πρέπει να είναι εκεί. Πρέπει να κατασβέσει την πυρκαγιά. Τελείωσε. Οι εθελοντές είναι επαγγελματίες και πρέπει και αυτοί να δουλέψουν σαν στρατός. Δεν είναι δουλειά ελεύθερης επιλογής αυτή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει και εκείνη από την πλευρά της να διερευνήσει όλα όσα πρέπει να εξεταστούν και να απαντηθούν. Γιατί αλλιώς θα αποθαρρυνθούν οι εθελοντές πυροσβέστες και δεν θα πηγαίνουν να βοηθούν τις κοινότητές τους και όταν προκύψει κάποια καταστροφή δεν θα υπάρχουν εθελοντές. Και τώρα με την κρίση δεν έχουμε την πολυτέλεια. Δεν, δεν, καλυπτόμεθα μόνο από τους ε, επαγγελματίες. Πρέπει οι θελοντές να αντιμετωπίζονται σωστά λοιπόν. Άρα θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα να εξεταστούν και να απαντηθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Μποστινάρου. Άλλος κανείς. Κανείς. Κανείς δεν ζητεί το λόγο. Λοιπόν, Α, θέλει τρία λεπτά ο αναφέρον. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Από αυτά που άκουσα, εάν εκτιμούμε τους εθελοντές, τους επαγγελματίες πυροσβέστες, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας την υγεία τους. Γιατί τελικά αυτοί οι άνθρωποι ε, δουλεύουν Ατελείωτε ώρε εργασία. Αν θέλουμε να του σεβαστούμε θα πρέπει να ανησυχήσουμε λοιπόν και για το χρόνο ανάπαυσής του. Η Ευρώπη λέει 48 ώρες. Ε, σε μια περίοδο αναφορά ε, τετράμινη. Ο υπολογισμό πρέπει να γίνει λαμβάνοντα υπόψη ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν και πλήρη απασχόληση. Ε, εδώ έχουμε στο Βέλγιο τον κανόνα των 38 ώρων. Δεν μου αρέσει να δίνονται παραδείγματα χρησιμοποιώντας το Βέλγιο έτσι, γιατί εδώ πέρα έχουμε 38 ώρες αντί 48. Ε, εγώ έκανα την παρέμβασή μου με βάση την ευρωπαϊκή νομοθεσία, την οποία πρέπει να σεβαζόμαστε. Εφόσον υπάρχει σχετική νομοθεσία, τη ζητάω να εφαρμοστεί, να εφαρμοστεί αυτό που είναι γραμμένο. Το θέμα δεν είναι αν δουλεύουν ή δουλεύουν. Ε, η απόφαση του δικαστηρίου με την απόφαση Αγκέρ λέει ότι το βασικό είναι που βρίσκονται. Δεν με ενδιαφέρει που είναι το Γέγκερ. Ε, υπάρχει μια διαφορά. Άλλο το σπίτι του πυροσβέστη και άλλος ο πυροσβεστικός σταθμός. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε το σπίτι του ως πυροσβεστικό σταθμό, ως παράτημα του πυροσβεστικού σταθμού. Έχουμε ένα υπουργικό ε, μια υπουργική εγκύκλιο που λέει πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Λέει, μπορείτε να είσαστε και εκτός του πυροσβεστικού σταθμού, μπορεί να είσαστε στο πιστρό, μπορεί να είσαστε στο καφέ. Δύο λεφτά όμως από το σταθμό ή πέντε λεφτά, έτσι λέει η Υπουργική η υπουργικη εγκυκλιος Τους περιορίζει. Επομένως το αίτημά μου είναι πολύ απλό. Αυτά που μου λέτε δεν θέλω να τα λάβω υπόψη μου όλα τα επιχείρηματά μου βασίζονται στις 48 ώρες που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Και είναι παλιά νομοθεσία. Θα ήθελα λοιπόν να την εφαρμόσουμε για τους ε, πυροσβέστες και τους καπανείς πυροσβέστες. Γιατί από αυτή την ε, νομοθεσία εξαρτάται, από... εξαρτάται η υγεία τους. Ένας ε, οδηγός, ας πούμε, φορτηγού πρέπει να σταματήσει ένα χρονικό διάστημα γιατί υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες αλλά ε, παρόλα αυτά επιβάλλεται ή μάλλον αφήνεται έναν πυροσβέστη αν χρειαστεί να πούμε να οδηγήσει όλη τη νύχτα. Δεν είναι σοβαρό αυτό. Ε, το Βέλγιο λέει ότι οι πυροσβέστες πρέπει να είναι έτοιμοι εντός 25 λεπτών. Φανταστείτε κάποιους άλλους, ας πούμε, να θέλουν μόνο 25 λεπτά για να κάνουν μια σοβαρή παρέμβαση η υπουργική μας εγκύκλειος λέει 2 ή 5 λεφτά. Είναι στο χώρο εργασία, στο χώρο εργασία τους. Είναι χρόνος εργασίας αυτός. Ναι. Εγώ δεν θέλω λοιπόν τίποτα άλλο παρά να σεβαστούμε την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Αφήστε το τι γίνεται στο Βέλγιο. Να ασχοληθούμε μόνο με το τι λέει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, που είστε τόσο ευγενικοί και με αφήσατε να καταχραστώ το χρόνο σας. Εγώ δεν είχα δει τη σχετική νομοθεσία. Σα ζητώ συγγνώμη. Γι' αυτό παίρνω το λόγο τώρα για να απαντήσω. Νομίζω ότι η Κομισιόν έδειξε ότι γνωρίζει πάρα πολύ καλά όλη αυτή την ιστορία. Ε, αυτό που καταγγέλλεται το ξέρει πολύ καλά από την παρέμβασή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι φάνηκε. Μας περιέγραψε πολύ λεπτομερώς όλα όσα είναι εν εξελίξη όλα τα διαβήματα που έχουν γίνει. Επομένω, πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτή αυτή την αναφορά, ούτω ώστε η Κομισιόν να ξεπεράσει τη φάση τη επαλήθευση. Περιμένουμε με ανυπομονησία το έγγραφο που μα υποσχεθήκατε και αναγγείλατε σήμερα. Και από αυτό το έγγραφο θα εξαρτηθεί τι θα κάνουμε μετά, αν θα υποβάλουμε περαιτέρω ερωτήματα ή θα κάνουμε και άλλα διαβήματα προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ούτω ή άλλω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε με μεγάλη επαγγελματικότητα. Μα περιγράψαμε κάθε λεπτομέρεια όλα τα βήματα που έχει κάνει. Κρατάμε λοιπόν και εμεί ανοιχτή αυτή την αναφορά και κλείνουμε αυτή τη στιγμή τη συζήτηση για αυτό το θέμα και στι 5.30 ακριβώ θα περάσουμε στη συνεδρίαση των συντονιστών.